Okay, colleagues, I'm getting started very Λοιπόν, αρχίζω νωρί γιατί ξέρω ότι πιέζει ο χρόνος. Έχουμε επίτροπο σήμερα, ο οποίος έχει μόνο τρία τέταρτα όταν θα έρθει. Έχετε το σχέδιο της ημερήσιας διάταξης ενώπιό σας. Εσείς οι τρεις που είστε παρόντες, είναι εγώ τέσσερις, συμφωνούμε εμείς οι τέσσερις. Το σχέδιο ημερήσιας διάταξης. Ωραία. Προχωρώ λοιπόν. Θέσπιση του προγράμματος Ορίζον 2020 εξέταση τροπολογιών, το λόγο έχει η κυρία Γκρισμπέκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Όσοι ήθιστε, ε, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω όλους τους κοιόδης συγγητές για τις άριστες ε, σχέσεις που είχαμε και την αγαστή συνεργασία τους τελευταίους μήνες για τη σύνταξη της έκθεσης. Με συμβαστικές τροπολογίες νομίζω καταφέραμε να συμπλησιάσουμε κάποιες απόψεις που δεν ήταν ε, προφανές αυτό και αυτονόητο από την αρχή γιατί μπορεί να έχουμε διαφορές για το ρόλο των ε, μεταφορών στην ευρωπαϊκή οικονομία και τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. Έχετε το κείμενο, το διαβάσατε φαντάζομαι και ποια είναι τα βασικά σημεία. Συμφωνούμε όλοι οι λίγοι παρόντες, σε πάση περιπτώσει, ότι θέλουμε να θεωρήσουμε τις μεταφορές στην Ευρώπη ως στοιχείο μεγέθυνσης οικονομίας, ανταγωνιστικότητας, αηφόρου ε, ανάπτυξης, ε, εδαφικής ε, συνοχής. Το τονίζουμε αυτό πάρα πολύ και βεβαίως σκεφτόμαστε και τι σημαίνει ως προς τις θέσεις εργασίας, τα κοινωνικά και τους γενικότερους στόχους για τις μεταφορές. προσθέτουμε επίσης και τις ανησυχίες και τα μελήματά μας για την ασφάλεια. Εκατό και κάτι είναι οι τροπολογίες που κατατέθησαν, τέσσερις συμβιβαστικές. Ε, ε, δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, απλώς να επανέλθω σύντομα στο ε, τι αναφέρουν. Η πρώτη συμβιβαστική είναι με τροπολογία της κυρίας Ντουιρόν που μιλάει για την αλλαγή των αναγκών ε, και των πολιτών. Ε, συμφωνούμε, μας έπεισε η κυρία Τυράν, ε, κυρίως για τις αστικές περιοχές. Γενικότερα, με το συμβασμό αυτό βρήκαμε μια αρκετά καλή ισορροπία ανάμεσα στην επιτακτική ανάγκη να μειωθούν οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα μαζί με την ανάγκη να μην περιθωριοποιούνται ακόμα περισσότερο οι ιδιαίτερα απομακρυσμένε περιφέρειες. Στη δεύτερη συμβιβαστική ε, έχουμε συνδυάσει πολλέ τροπολογίε ε, που αναφέρονται στη σημασία των μεταφορών στην Ένωση διότι ε, δημιουργούν θέσεις εργασίας, πάνω από 13 εκατομμύρια θέσεις εργασίας, αν δεν με πατάει η μνήμη μου, και αυτό είναι σημαντικό στο κοινοτικό ΑΕΠ, πάνω από 6% και έρχεται εδώ να προσθεθεί βεβαίως και η ενέφτη της εδαφικής ε, συνοχής. Η αρχική τροπολογία ε, είχε αντικαταστήσει τροπολογία 56 της κυρίας Ντεβεράκ που μιλούσε για ανάκαμψη της οικονομίας και της ε, βιομηχανίας και τόνιζε την αεροναυπηγική που είναι σημαντικός μοχλός στην Ένωση και παραμένει και τελικά κάνω μια συμβαστική αλλά διαφώνησε το ΕΛΚ. Και τελικά ε, αποσύρθηκε η τροπολογία 56 από το συμβασμό και θα ψηφιστεί χωριστά. Ε, για την τρίτη συμβαστική τροπολογία που είναι η ίδια η ουσία της ε, έκθεσης έρευνα και καινοτομία τονίζεται η ανάγκη να μειωθούν οι εκπομπές ε, διοξιδίου του άνθρακα 2020-2050 και επίσης τονίζουμε τη σημασία να μειωθούν στο μισό τα θύματα από τροχέα ε, στους αυτοκινητοδρόμους μας μέχρι το 2020. Αυτό το θυμήσαμε και το ψηφίσαμε και στην έκθεση ΚΟΧ με στόχο να ε, έχουμε μηδέν θύματα στην άσφαλτο μέχρι το 2050. Αυτά. Οι άλλες αλλαγές είναι λίγο ε, διακοσμητικές. Στα γαλλικά αλλάξαμε ε, το ρήμα conduit και βάλαμε des. Στα γαλλικά δεν αλλάζει πάρα πολλά πράγματα, αλλά στα αγγλικά άλλο είναι το βοηθά και άλλο ε, οφείλει να οδηγεί. Ένα τελευταίο για την τελευταία συμβαστική τροπολογία. Σημαντική μείωση του διοξιδίου του άνθρακα, είπαμε, των εκπομπών και αυτή η στόχη Περνώ από τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης όλων των μέσων μεταφοράς, χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, το σιδηρόδρομο, στις ναυτικές, ναυτιλιακές μεταφορές και στις αερομεταφορές και τελικά ε, προτείνουμε να συμπεριληφθούν και τα όσα έχουμε εκπονήσει για τα εναλλακτικά και φορά καύσιμα, αλλά και ε, συστήματα προώθησης νοτόμα αποτελεσματικά και βελτιστοποίηση των συστημάτων ε, τροφοδοσίας στο καύσιμο. Και θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη και ε, το βάρος των αυτοκινήτων και η αεροδυναμική τους στην κατασκευή των αυτοκινητοδρόμων. Επισυνάφτεται ο κατάλογος ψηφοφορίας για τις 100 και πλέον τροπολογίες. Κάνω κάποιες προτάσεις ε, για ορισμένες τροπολογίες. Ε, λέγω ότι είμαι αντίθετο, όχι γιατί είναι κακές χαμηλότερης ποιότητας, αλλά μαζί με τους κοιόδης ηγητές θελήσαμε να είμαστε ιδιαίτερα στοχευμένοι στην έκθεσή μας ε, με κέντρο βάρου στην έρευνα και την καινοτομία, γιατί αυτό ε, μας ζητούσε και ο τίτλος της έκθεσης. Και δεν θέλαμε να την αποδυναμώσουμε επαναλαμβάνοντας κάποια πράγματα που έχουμε ήδη πει αλλού. Επίσης, προτείνω να μην γίνει δεκτή η τροπολογία 71 της κυρίας Ντυρό που μιλά για την πράσινη φοδιαστική. Πολύ ενδιαφέρουσα έννοια αυτή, αλλά δεν έχει καμία σχέση εδώ με την έρευνα και την καινοτομία. Και περιτεύει το ίδιο για την τροπολογία 99 ε, της κυρίας Αγιάλα Σέντερ. Μπορεί να χρειάζεται συμμετοχή του κοινού, διαβούλευση ε, στη χάραξη των μεγάλων αξώνων υποδομών και των μεγάλων έργων, αλλά αυτή η τροπολογία ανήκει στην έκθεση για τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών και όχι σε αυτή εδώ. Αυτά τα βασικότερα με στη διάθεσή σας αγαπητοί συνάδελφοι, αύριο το πρωί ψηφίζουμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Thank you very much, Mr. Ευχαριστώ, ο κύριος Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ο σκιώδης εισηγητής μας δεν έχει έρθει ακόμα, γι' αυτό στο όνομα του ΕΛΚ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την πολύ καλή δουλειά που έχει κάνει ε, διότι στα θέματα αυτά κινδυνεύει κανείς ε, συχνά να θέλει να τα πει όλα και να ε, μην λέει τίποτα τελικά. Νομίζω ότι αυτό δεν συμβαίνει στην περίπτωση αυτή σε μια πολύ καλή συζήτηση με τις άλλες πολιτικές ομάδες νομίζω ότι έχει υπογραμμίσει τα σωστά σημεία. Στην Επιτροπή μας έχουμε πει ότι το Κοινοβούλιο αλλά και η Κομισιόν θα πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι γενικά στην στρατηγική 2020 και ιδιαίτερα όσον αφορά την έρευνα και την ανάπτυξη η κινητικότητα και οι μεταφορές μπορούν να αποτελέσουν πολύ σημαντικό εταίρο ο οποίος πολύ συχνά υποτιμείται ε, και όσον αφορά την οικονομική αξία και όσον αφορά την ε, δυνατότητα να ενισχύσει τις ε, έρευνες ε, στην Ευρώπη. Στην έκθεση νομίζω ότι αυτό παρουσιάζεται σωστά και γίνονται πολύ σωστά γεφυρώματα ανάμεσα στην, στις μεταφορές και στην κινητικότητα ως οικονομικό παράγοντα αλλά και στις προκλήσεις όσον αφορά την βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτά είναι περισσότερο από αυτονόητα για μας ε, και επίσης ε, θα ήθελα να εκφράσω την κατανόησή μου για την ε, τροπολογία της Κριστίν Ντεβεράτ όσον αφορά τις αερομεταφορές, διότι για μένα αυτό είναι ένα από τα βασικά παραδείγματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο όπου έχουμε συνεργαστεί ε, οι χώρες μεταξύ μας ε, και μπορώ να φανταστώ ότι ακόμα και οι πράσινοι, αγαπητέ Μίχαελ, ε, θα ξεπεράσουν τον εαυτό τους και θα θεωρήσουν αυτή την πρόκληση σε ευρωπαϊκό επίπεδο παράδειγμα για να πούν ότι αυτή την συνεργασία την θέλουμε και σε άλλους τομείς. Ίσως μπορούμε να γυρίσουμε την τροπολογία έτσι ώστε να την υποστηρίξουν όλες οι πολιτικές ομάδες. Εμείς στηρίζουμε την ε, έκθεση, στηρίζουμε και ε, τις τροπολογίες αυτές ε, με τις αποχρώσεις που τονίζουν ποια είναι η πραγματικότητα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κράμερ. Η σκιώδηση συγκήτριά μα ε, δεν έχει έρθει ακόμα, γι' αυτό θα ήθελα στο όνομά τη να ευχαριστήσω την ε, εισηγήτρια. Ε, στηρίζουμε τις ε, συμβαστικές τροπολογίες που έχουν υποβληθεί, αλλά όσον αφορά ε, το σημείο που ανέφερες, δεν υπάρχει συμβαστική τροπολογία, δεν μπορούμε λοιπόν να τη στηρίξουμε. Είμαστε υπέρ της διασνορικής συνεργασίας και της ευρωπαϊκής διάστασης, όχι μόνο σε αερομεταφορές, γενικά και στις έρευνας, αλλά δυστυχώς δεν μπορέσαμε να καταλήξουμε σε ένα συμβιβασμό. Γι' αυτό οι πράσινοι θα πρέπει να καταψηφίσουν. Ματιέ, όμως νομίζω ότι το ε, Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Φώστερ. Thank you very much, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ την ε, Ναταλή Γκρισμπερ για την ασκλή δουλειά τη. Είναι πολύ περίπλοκη η έκθεση. Ζητώ συγγνώμη εξ ονόματο του σκιώδου εισηγητού μα, του κύριου Σίζων. Ε, δεν είναι εδώ. Όλοι εξετάζουμε τον κατάλογο ψηφοφορία πολλά πράγματα μπορούμε να τα υποστηρίξουμε από πλευρά τη ομάδα μα. Υπάρχουν βεβαίω κάποια ερωτήματα, αλλά ευχαριστούμε τον εισηγητή ακόμα μια φορά, την εισηγήτρια μάλλον, για τη δουλειά τη. Η κυρία Γιάλα Σέντερ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για αυτή την έκθεση αναγνωρίζω τις καλές προθέσεις ε, της κυρίας Δεβεράκ με αυτή την έκθεση. Θέλω να πω ότι όντως η αεροπορία ε, χρειάζεται πολύ έρευνα, αλλά και οι άλλοι τομεί το ίδιο. Δεν μπορούμε να μιλάμε μόνο για την αεροπορία. Γι' αυτό ακριβώς εγώ θα προτείνω μια προφορική τροπολογία. Ε, θα πρέπει να υπάρξουν περισσότερε ευρωπαϊκέ δεσμεύσει για όλου του τομεί μεταφορών, ε, δεδομένη τη οικονομική του σημασία. Γιατί πραγματικά όλοι οι τομεί ε, έχουν ανάγκη ε, περισσότερη έρευνα. Ε, δεν διαφωνώ σε καμία περίπτωση με την αεροπορία, με το να υποστηρίξουμε την αεροπορία, αλλά και άλλοι τομεί χρειάζονται υποστήριξη όπω και η αεροπορία. Δεν πρέπει λοιπόν να προωθούμε εμεί αυτέ τι διακρίσει μόνο υπέρ τη αεροπορία. Ευχαριστώ. Η Κομισιόν. Ο κύριος Νταμιάννη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Από πλευράς Κομισιόν, μπορούμε να πούμε ότι μας άρεσε η έκθεση της εισηγήτριας. Μέσα σε ένα επικοδομητικό πνεύμα συζητήσαμε και μαζί της αλλά και με την υπόλοιπη Επιτροπή και τα μέλη της. Η έκθεσή της δικατοπτρίζει ε, την πραγματική έννοια, τον πυρήνα, αν θέλετε, της πρότασης της Κομισιόν ορίζοντας 2020. Και ειδικά το τμήμα που αφορά τις μεταφορές. Προσπαθήσαμε να έχουμε μια ισορροπία ανάμεσα στην υποστήριξη των πολιτικών, την οικονομική και βιομηχανική ανάπτυξη, με στόχους που προωθούν την τεχνολογία Θέλουμε δηλαδή και μια οριζόντια μεταφορά, οριζόντια αντιμετώπιση των μεταφορών από τη μία, αλλά να αναγνωρίσουμε και τις ιδιαιτερότητες του κάθε τρόπου μεταφοράς όταν χρειάζεται. Η εισηγήτρια έδωσε έμφαση και ορισμένε από τις τροπολογίες επίσης που πρότειναν και οι άλλοι ευρωβουλευτές έδωσαν έμφαση την ανάγκη να ενισχύσουμε τις σχέσεις με τις σχετικές πολιτικές. Πολύ καλή ιδέα. Όχι μόνο με την πολιτική μεταφορών, αλλά πολιτική κλίματος, ε, περιβάλλοντος και ενέργειας, οι στόχοι της πολιτικής όπως λέμε. Επίσης, να ενισχύσουμε τη συμπληρωματικότητα με άλλα προγράμματα και άλλα τμήματα του ίδιου προγράμματος. Και επιπλέον έμφαση στην αηφορία επίσης δίδεται. Αυτό τι σημαίνει. Για όλους αυτούς τους λόγους είμαστε υπέρ πολλών τροπολογιών που προτείνονται. Τώρα, υπάρχουν κάποιες άλλες που δεν μας βρίσκουν τόσο σύμφωνους βέβαια. Κυρίως αυτές οι τροπολογίες που εισαγάγουν ένα υπερβολικό επίπεδο λεπτομέρειας. Μερικές φορές προσπαθούν να παντρέψουν ε, διάφορες ιδέες. Ε, προσπαθείτε εσείς επίσης να προτείνετε συμβιβαστικές τροπολογίες, αλλά εκεί υπάρχουν μερικές αντιφάσεις. Παραδείγματο χάρη συμβαστική τροπολογία 4 έχει τέτοιες αντιφάσεις. Oh. Σε κάποιες περιπτώσεις που καταβάλλεται μια προσπάθεια με ΑΙ να μπουν κάποια στοιχεία που είναι εκτός του βασικού πεδίου της πολιτικής μεταφορών. Παραδείγματο χάρη η εισαγωγή του τουρισμού. Συνολικά πάντως μπορώ να πω ότι είμαστε πολύ θετικοί και είμαστε υπέρ πολλών τροπολογιών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η εισηγήτρια θέλει να προσθέσει κάτι. Μετά από τόσους επένους της Κομισιόν, μπορεί κάτι να θέλετε να πείτε. Τι να πω, δεν θέλω να προσθέσω τίποτα. Ε, Έμεινα με ανοιχτό στόμα από τους τόσους επένους με τους οποίους με έρανε η Κομισιόν. Πώς συνέβη αυτό. Διερωτώ με. Όχι, όχι, αστείο ήταν αυτό. Χαίρομαι που συμφωνούν πάρα πολύ με τη δουλειά μου και συμφωνώ με την Κομισιόν ότι όντως είναι πιο απλό να προσπαθήσουμε να επικεντρωθούμε καλύτερα, να είμαστε πιο ε, λακωνικοί και για να και για να αποφύγουμε και τις αντιφάσεις, έτσι. Ακριβώς γι' αυτό κάναμε αυτέ τις συμβαστικέ τροπολογίε εξάλλου. Καταλαβαίνω επίση αυτό που είπε για την ε, συμβαστική τροπολογία 4, αλλά έτσι γίνεται με αυτέ τι ε, προσπάθειε. Προσπαθούμε να βρούμε ισορροπία με τέτοιου συμβασμού. Άκουσα επίση την πρόταση για προφορική τροπολογία τη Ινέσα Γιάλα Σέντερ. Την υποστηρίζω απόλυτα. Είναι μια θαυμάσια ιδέα. Σε ό,τι αφορά τώρα τις παρατηρήσεις του Ματιέ Γκρός, του Μίκαελ Κρέμερ και της κυρίας Φώστερ, συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπαν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα ψηφίσουμε αύριο. Να υπενθυμίσω ότι ψηφίζουμε στην Επιτροπή Ήτρε τον Οκτώβριο και θα περάσει στην Ολομέλεια του Νοεμβρίου. Καταρχήν, έτσι. Γιατί ξέρετε πολύ καλά τι γίνεται με τους οροφές ε, της ε, Ολομέλειας, οπότε μπορεί να αλλάξουν και οι μερίσεις διατάξεις της Ολομέλειας. Πάμε τώρα στα δικαιώματα των επιβατών ε, σε όλους τους τρόπους μεταφοράς. Ο εισηγητής είναι ο κύριος George Bach. Έχεις το λόγο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους συναδελφούς για τις ιδέες τους που ε, μεταφράζεται σε 250 τροπολογίες παρακαλώ. Και είμαι βέβαιος ότι δεν μας χωρίζουν μεγάλες πολιτικές διαφορές. Αν κοιτάξετε τις διάφορες προτάσεις, διαπιστώνετε ότι περισσότεροι συνάδελφοι ζητούν περισσότερο από τον εισηγητή και ε, έχουν προτείνει νέες ιδέες που εμπλουτίζουν και συμπληρώνουν την έκθεση. 12 συμβιβαστικές προτείνουμε και αυτές επικεντρώνονται στα βασικότερα σημεία όπως είναι η διαφάνεια, η πληροφόρηση, η πρόσβαση για άτομα με αναπηρίες και περιορισμένη κινητικότητα και επίσης διαδικασίες καταγγελιών και παραπώνων. Και στο θέμα της αφαιρεγγιότητας ε, αεροπορικών εταιριών είναι και επίκαιρο. Έχουν γίνει πολλές τροπολογίες ε, πέρα από διάφορες ε, πολιτικές ομάδες και από τις δικές μου προτάσεις προτείνουν περισσότερα. Γι' αυτό για να ανταποκριθούμε σε αυτά τα αιτήματα έγινε μια πολύ φιλόδοξη ε, συμβαστική τροπολογία για να προστατεύονται οι επιβάτες απέναντι σε τέτοια δυσάρεστα φαινόμενα και δυσάρεστες συνέπειες. Θα το συζητήσουμε. Ξέρουμε τι ζητάει ο κλάδος και Περιμένω με αγωνία και ενδιαφέρον να ακούσω τι θα πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά. Έχουμε και ψήφισμα του Κοινοβουλίου του 2009, αλλά έκτοτε δεν έχουν ληφθεί καθόλου μέτρα. Ήδη από το 2009 το Κοινοβούλιο ζητάει σαφή ε, λήψη θέσης. Ε, βεβαίως προσπάθησα τις περισσότερες προτάσεις σας ε, να τις εγκρίνω στον κατάλογο ψηφοφορίες να βάλω ένα συν δίπλα. Δυστυχώς καμιά φορά χρειάστηκε βάλω και αρνητικό ε, πρόσημο. Γιατί και η λογική και η συνέπεια το επέβαλα. Οι συνάδελφοι σάφησα και Ουτίας πρότειναν να λάβουμε υπόψη μας και τους ηλικιωμένους που δεν ξέρουν πάντα όλες τις σύγχρονες τεχνολογίες όταν ταξιδεύουν. Αυτό δεν έχει να κάνει με την ηλικία. Γιατί οι πιο ηλικιωμένοι. Υπάρχουν ηλικιωμένοι που είναι σαΐνια στις τεχνολογίες, ενώ κάποιοι νεότεροι που δεν τα πάνε και τόσο καλά. Και πώς θα τους λάβει υπόψη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο συνάδελφος Τρέιλερ έχει κάνει ε, πολλές προτάσεις που καλούνται οι εθνικές ε, αρχές να γίνουν ανεξάρτητες αρχές, να αλλάξει διατύπωση. Καταλαβαίνω ε, καταρχήν τι θέλει, αλλά οι εθνικές ε, εφαρμοστικές αρχές είναι κάτι το οποίο υπάρχει στα αγγλικά σε όλες τις νομοθετικές προτάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα το βρείτε και αλλού. Γι' αυτό, για λόγους απλούστευσης προτείνω να ε, καταψηφίσουμε αυτή την τροπολογία. Επίσης θα παρακολουθώ τον κύριο Τέιλορ να μου πει κάτι για την 176 τροπολογία του για τους παρόχους ε, υπηρεσιών ε, που μιλάει για την αφαιρεγκαιότητα. δηλαδή τι είναι, δεν είναι μόνο οι αεροπορικές εταιρείες, ποιους άλλους εννοεί. Επίσης, οι συνάδελφοι Τρεμόσα, ε, Βλάστο, Ντεβεράκ, ε, και άλλοι και η κυρία Σάβιζα αναφέρονται στο overbooking και στο overselling. Ε, ίσως θα μπορούσαμε να μάθουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά πόσο το έχει κοιτάξει και καλύπτεται από τις νομοθετικές προτάσεις που πρόκειται να μας υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χρειάζεται ιδιαίτερη μνήα. ένα τυπικό στο τέλος. Κατανοώ τα επιχειρήματα κάποιων συναδέλφων που εξάφρασαν παράπονα ότι δεν είχαμε χρόνο για να ε, συζητήσουμε τα θέματα σε μεγάλο βάθος. Και εγώ θα ήθελα να έχω περισσότερο χρόνο. Αλλά ε, είχαμε πρόβλημα με τις μεταφράσεις που τις ε, πήραμε την περασμένη εβδομάδα που ήταν εβδομάδα Στρασβούργου που δεν έχουμε χρόνο έτσι κι αλλιώς να κάνουμε τέτοιες τεχνικές συνεδριάσεις αλλά ζητώ οπωσδήποτε το Κοινοβούλιο στην Ολομέλεια ε, τον Οκτώβριο να ψηφίσει. Αν θέλουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συμπεριλάβει ε, τις εργασίες της, Αυτό που θα πούμε εμείς για τους επιβάτες ε, των αεροπορικών εταιριών, γιατί το Νοέμβριο θα φέρει την πρότασή της. Ήθελα να σας πω ότι στα τέλη της περασμένης εβδομάδας ε, Αφαιρέθηκε η έκθεση αυτή από τη Σύνοδο του Οκτωβρίου μαζί με άλλα θέματα. Για τους λόγους που σας ανέφερα θα ήθελα όμως να παρακαλέσω τους συντονιστές να ε, ασκήσουν πίεση στην πολιτική του ομάδα ο καθένας για να επανέλθει στην ημερήσια διάταξη το θέμα και όπως είχε προβλεφθεί και όπως επιβάλλει η τάξη να ψηφιστεί τον Οκτώβριο. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Κύριε Μπαχ, να επαναλάβω το τελευταίο θέμα για τους συντονιστές. Να έρθουν σε επαφή με τους συντονιστές, για να... οι οποίοι μπορούν να επευθυνθούν συνεχεία στους πολιτικούς ηγέτες για να επανέλθει το θέμα στη μερίσια διάταξη. Ο κύριος Γκρός έχει ήδη ασχοληθεί και ο κύριος Ντο... και οι υπόλοιποι τέλο πάντων, ο κύριος Αλκαντράουι, Μάικλ και εσύ, να έρθει σε επαφή με τους αρχηγούς των ομάδων σας να έρθετε σε επαφή με τους αρχηγούς των πολιτικών ομάδων σας για να επανέλθει το θέμα στη μερική διάταξη. Ξέρουμε ότι έχουμε πρόβλημα με τα ταβάνια. Αλλά μπορεί τελικά εμείς να ετοιμάσουμε την έκθεσή μας μετά την Κομισιόν. Δεν είναι ακριβώ αυτό που θέλουμε, έτσι. Λοιπόν, από τους σοσιαλιστές τώρα η σκιώδη συγγήτρια. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την ε, και καλή του θέληση και την καλή δουλειά του. Ε, μπορούμε να υποστρίξουμε την έκθεση με μικρές αλλαγές. Συμφωνώ με αυτά που υπόθηκαν προηγουμένως ότι είναι πολύ σημαντικό να στείλουμε ένα μήνυμα στην Κομισιόν εγκαίρως πριν ετοιμάσει και εισαγάγει την πρότασή της. Ε, δουλέψαμε εμείς πραγματικά έντονα. Προσπαθήσαμε τον εισηγητή να είμαστε πολύ ε, επικοδομητικοί και συμφωνούμε με τη συμβαστική τροπολογία Β, να δημιουργήσουμε δηλαδή ένα κοινό νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη και τις ιδιαιτερότητες των διαφόρων ειδών μεταφορών, αλλά και θα έχει και μια οριζόντια θεώρηση των πραγμάτων. Σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των δικαιωμάτων των επιβατών, τώρα για την αφαιρεγκαιότητα και την προστασία των πελατών των επιβατών δηλαδή. Είναι πολύ σημαντική για αυτό το θέμα η τροπολογία 8. Ιδίω για του επιβάτε που έχουν μειωμένη κινητικότητα. Θα πρέπει να έχουμε και υπηρεσίε βοήθεια. Επίσης, ε, η πολιτική τιμών θα πρέπει να διαφανείς, η πληροφορία θα πρέπει να δίδεται με πολύ φιλικό τρόπο, σε διάφορες γλώσσες, να είναι εύκολα προσπελάσιμη. Επίσης, για τις πληροφορίες. Δεν θέλουμε περίπλοκα συστήματα. Σύντομες πληροφορίες ή τα δικαιώματα των επιβατών στα εισιτήρια πρέπει να αναγράφονται. Μπορούμε να υποστηρίξουμε σαφέστατα την έκθεση με κάποιες μικρές λεπτομέρειες που πρέπει να ξαναδούμε. Αλλά επαναλαμβάνω ακόμη μια φορά, ευχαριστώ τον εισηγητή για την συνεργασία του. Κύριε Σαβισάρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Είναι μια έκθεση πρωτοβουλίας και πρέπει να έχουμε μια πολύ συγκεκριμένη θέση απέναντι στο κείμενο της Κομισιόν. Ευχαριστώ τον εισηγητή για την πρότασή του. Σε αυτή την έκθεση παρουσιάσαμε τελικά πολύ λίγες τροπολογίες. Η πλειοψηφία των συναδέλφων αναφέρθηκαν σε αυτή την ανησυχία που είχαν για, τις, για τα δικαιώματα των επιβατών. Γι' αυτό ακριβώς κάναμε κάποιες τροπολογίε, οι οποίες γενικά την χάνουν υποστήριξη. Και στηρίζουμε τη θέση του εισηγητή σε σχέση με τις προτάσεις της Επιτροπής ΣΥΜΚΟ. Δεν υπάρχει λόγος να μπω σε λεπτομέρειε. Μία ερώτηση έχω να κάνω μόνο. για τις τροπολογίες 60 και 62, σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στις πληροφορίες. Ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει τεχνολογία, όλοι τη χρησιμοποιούμε πολύ. Φυσικά όλοι θα πρέπει να χρησιμοποιούν τα smartphones, τα έξυπνα τηλέφωνα. Θα πρέπει να είναι σε θέση να τα χρησιμοποιήσουν. Υπάρχουν όμως άνθρωποι που δεν έχουν κινητά τηλέφωνα. Υπάρχουν και αυτοί ή που δεν χρησιμοποιούν ε, το ίντερνετ. Και καμιά φορά είναι ηλικιωμένοι. Ε, να μην τους ξεχνάμε και αυτούς, να λάβουμε υπόψη τις ανάγκες τους. Πώς μπορούμε να τους ε, συμπεριλάβουμε στην έκθεση, πώς μπορούμε να τους δώσουμε τις πληροφορίες που χρειάζονται αυτά τα άτομα. Θα πρέπει και αυτοί να μπορούν να πληροφορούνται ό,τι χρειάζονται χωρίς να πρέπει να έχουν και καλά κινητά. Η τροπολογία που αφορά την πρόσβαση των πληροφοριών. Εντάξει, υπάρχουν οι νέες τεχνολογίες και εδώ. Μερικά όμως άτομα ε, πρέπει να τα βοηθήσουμε, ε, να τα καταρτήσουμε, ώστε να βοηθήσουν τους υπόλοιπους που δεν έχουν εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες. Επίσης, ε, οι επιβάτες ορισμένων, σε ορισμένες περιοχές ε, αναγνωρίζουν, αντιμετωπίζουν δυσκολίες για συγκεκριμένους λόγους. Εδώ θα πρέπει να έχουμε τα κατάλληλα συστήματα, ούτως ώστε να μην ξεχνάμε κάποιους επιβάτες, να μην τους παρατάμε αυτό το πρόβλημα. Επίσης, για το overbooking και overselling. Μην ξεχνάμε και εδώ ότι πρέπει να έχουμε σαφείς κανόνες για τους επιβάτες. Αυτά είναι κάποια επιμέρους σχόλια, αλλά γενικά υποστηρίζω την έκθεση. Ο κύριος... Ευχαριστώ πολύ, ο κύριος Κράμερ. Να ευχαριστήσω και εγώ τον εισηγητή ε, για την ε, καλή συνεργασία και την καλή έκθεση. Στηρίζουμε τη συμβαστική πρόταση και την έκθεση αποφασιστική σημασία για μας είναι να υπάρχει ένα ε, ανεξάρτητο κέντρο διαιτησίας για όλα τα είδη μεταφορών. Οι αερομεταφορές ήταν κατά, οι σιδηρόδρομοι ήταν υπέρ και οι περισσότερες περιπτώσεις λύνονται συνενετικά. Ε, σε πτήση της Brussels Airways. Ε, εμένα μου έκανε εντύπωση ότι είχα καθυστέρηση. Ε, ρώτησα γιατί δεν μπορούσαν να μου πούνε. Τους είπα ότι θέλω αποζημίωση. Δεν μου δεν μου έδωσαν ε, και ε, έφτασα στη πύλη και μου είπαν ότι ακυρώθηκε η πτήση και ε, έκανα παράπονα και με αποζημίωσαν, αλλά μάλλον επειδή είμαι ευρωβουλευτής. Τι γίνεται σε περίπτωση που παραβιάζονται οι κανόνες που υπάρχουν. Αυτή είναι η ερώτησή μου προς την Επιτροπή. Μία ομάδα ήταν στην Ιταλία, ακυρώθηκε ένα τρένο Πρώτα είχαν είχαν ανά πέντε λεπτά. Μετά από δύο ώρες είπαν ότι ακυρώνεται η διαδρομή. Ε, και φτάσανε, αυτό ήταν τρένο Intercity με το τελευταίο περιφερειακό τρένο τελικά. Ε, ε στο, τρένο αυτό ήρθε ο ε, ελεγκτής και τους ε, έδιωξε από το τρένο επειδή είπε ότι δεν ισχύει το ε, εισιτήριο και ήρθε η αστυνομία και του ε, κατέβασε από το τρένο. Αυτό είναι το τελευταίο που χρειαζόμαστε, τέτοια εθνικιστική πολιτική του χείρις του είδου. Ε, και ε, θέλω να ρωτήσω, η Κομισιόν πώς θα παρέμβει, ποιο θα τιμωρείται και ακριβώς γι' αυτό δημιουργούμε αυτού τους κανόνες, θα πρέπει όμως να τηρούνται και γι' αυτό θα ήθελα από την Επιτροπή απάντηση. Θα μπορούσα να σα δώσω, να σας δείξω και άλλες επιστολές που μου στέλνουν ε, δεν επιτρέπεται ε, αυτά να περνάνε ατιμόρυτα. Λέει ο, ο, πελάτης έχει πάντα δίκιο, αλλά αυτό δεν το βλέπουμε στις περιπτώσεις αυτές, ε, στις μεταφορές. Και ε, όχι μόνο όταν πιάνει φωτιά ένα πλοίο που συζητήσαμε στην προηγούμενη συνεδρίαση, τι γίνεται και στην περίπτωση που για παράδειγμα κατεβάζονται από το τρένο επιβάτες επειδή ακυρώθηκε το κανονικό στο τρένο. Ε, ευχαριστώ κύριο Σάμπολ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εισαγωγικά θα ήθελα ε, να σχολιάσω το εξή. Ε, θα ήθελα να, να πω ότι χαίρομαι που ακούω ότι ο, ο κύριο Κράμερ έχει προβλήματα με την Brussels Airlines, διότι νόμιζα ότι μόνο εγώ έχω τέτοια προβλήματα, αλλά από ό,τι φαίνεται όχι. Και συμφωνώ όσον αφορά την έλλειψη πληροφόρηση που παρέχεται σε τέτοιε περιπτώσει. Κύριε Πρόεδρε, μια γενική παρατήρηση. Ήθελα καταρχήν να πω ότι όσον αφορά τις ε, τροπολογίες ε, που έχουμε και τις συμβαστικές προτάσεις, ε, είμαι υπέρ αυτών που γενικά είναι αναλογικές. Αυτό που θα πρέπει να αποφύγουμε είναι να είμαστε υπερβολικοί όσον αφορά τη δημιουργία γραφειοκρατικών προβλημάτων για τις επιχειρήσεις. Θέλουμε να προστατεύσουμε τους ε, επιβάτες, αλλά δεν θα πρέπει να, ε, να επιβάλλουμε υπερβολικό άχθο σε μικρές επιχειρήσεις. Ε, τούτου λεχθέντος ε, θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις σχετικά με τις ε, τροπολογίες. Γενικά, αρκετέ από τις συμβαστικές τροπολογίες αξίζουν την υποστήριξή μας, ιδιαίτερα αυτές που έχουν να κάνουν με την διαφάνεια Ε, ιδιαίτερα πιστεύω ότι οι συμβαστικές προτάσεις 1, 3, 6 και 7 είναι χρήσιμες. Ε, πολύ ευχαρίστως θα υποστηρίξω και την ε, τροπολογία 5 που θέλει να διασφαλίσει την ε, διαφάνεια κατά την ε, τιμολόγηση. Όσον αφορά τις συμβαστικές τροπολογίες 8 και 9, ε, νομίζω ότι εδώ έχουμε ένα πολύ βασικό θέμα όσον αφορά την προστασία των ε, επιβατών σε περιπτώσεις ε, αφαιρεγγιότητας. Το άλλο θέμα που θα ήθελα να θίξω έχει να κάνει με ε, τα άτομα με αναπηρίες και πολύ ευχαρίστω θα υποστηρίξω την ε, συμβαστική ε, τροπολογία 10 και επιτρέψτε μου κύριε Πρόεδρε να, να προωθήσω και τη δική μου τροπολογία την 20 που έχει να κάνει με τις προσαρμογές σε περιπτώσεις ε, επιβατών με σοβαρές αναπηρίες. Ελπίζω ότι οι συνάδελφοι θα υποστηρίξουν αυτή την τροπολογία. Θα ήθελα επίσης να συμφωνήσω με τον ε, κύριο Μπαχ και ε, όσον αφορά την παροχή πληροφοριών σε διάφορες μορφές. Εγώ δεν τα ε, καταφέρνω πολύ καλά με την ε, τροπολογία. Δεν έχω ούτε iPhone, ούτε iPad, ούτε τίποτα με i. Ε, εγώ θα ήθελα να τα έχω άσπρο μαύρο, σε χαρτί δηλαδή. Και είμαι βέβαιος ότι και άλλοι νεότεροι ή πιο ηλικιωμένοι από μένα θα εκτιμούσαν κάτι τέτοιο. Δεν κουβαλάμε όλοι καλά και γεμάτα από συσκευέ μαζί μα. Πάντως, γενικά, κύριε Πρόεδρε, στηρίζω την ε, την ε, πρόταση αυτή και θα ήθελα να ε, την υπερψηφίσει η Επιτροπή μας. Ο κύριος Κρόσε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όσον αφορά τα δικαιώματα των επιβατών είναι κάτι που μας έχει ξανααπασχολήσει και περνάμε... Έχουμε φτάσει σε κρίσιμη φάση με τον φάκελο αυτό και πρέπει να φροντίσουμε ε, να διεξάγουμε τη συζήτηση στο Κοινοβούλιο προτού να υποβάλει η Κομισιόν την ε, επόμενη της πρόταση. Από τις εμπειρίες που έχουμε από το παρελθόν θα ήθελα να συμφωνήσω με τους συναδέρφους που τονίζουν ότι πρέπει να έχουμε νομοθεσία που να είναι τόσο σαφής ώστε να μην ε, δίνει αφορμή για προσφυγές. Ε, ψάχνοντας να βρούμε παραθυράκια στην ομοθεσία και εξετάζοντας ε, τις ε, λεπτομέρειες, πολύ συχνά γίνονται τα πράγματα πολύ πολύπλοκα και δεν ξέρουμε πού ξεκινάνε τα δικαιώματα και πού τελειώνουν. Μπορούμε πολύ απλά να εκφράσουμε αυτό που έχουμε εκφράσει και σε άλλους τομείς, ότι πρέπει να έχουμε σαφείς συνομιλητές στα κράτη-μέλη και αυτοί οι συνομιλητές να έχουν τις ίδιες δυνατότητες. Τους ανθρώπους, ε, τους ενδιαφερόμενους δηλαδή, να μπορούν να τους απαντήσουν ε, στη γλώσσα τους. Ε, σε κάποιες χώρες είναι δύσκολο να λάβει κανείς πληροφορίες για γλωσσικούς λόγους. Και όχι στι περιπτώσει όπου έχουμε μια μικρή καθυστέρηση, αλλά σε σοβαρέ περιπτώσει θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα οι πληροφορίε ε, να δίδονται σε όλου του επιβάτε ε, εν μέρει στη μητρική του γλώσσα. Αυτό κατά τη γνώμη μου είναι πολύ σημαντικό. Η τελευταία παρατήρηση είναι η εκ των προτέρων ε, πληροφόρηση. Δεν θέλω να αναφέρω συγκεκριμένε αεροπορικέ εταιρείε, τι γνωρίζουμε όλες, όλοι, αλλά όταν κάνω μια κράτηση και λαμβάνω 12 σελίδες ε, με ένα σωρό πτυχές, πληροφορίες, ε, προθεσμίες, ε, προθεσμίες μετά τις οποίες να χάνω όλα μου τα δικαιώματα λίγο πολύ. Εκεί θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν τρεις-τέσσερις βασικές πληροφορίες που θα πρέπει να παρέχονται. Ε, ξέρω και τις επιγραμμικές ε, κρατήσεις όπου με ένα απλό κλικ ε, λέει κανείς ότι δέχεται όλα τα, όλους τους όρους αλλά δεν θα πρέπει να είναι τόσο πολύπλοκοι οι όροι θα πρέπει σε μια σελίδα να μπορούν να παρουσιαστούν Ζόρς νομίζω ότι δεν χρειάζεται να είναι τόσο πολύπλοκη η έκθεση αυτή νομίζω Ζόρς ότι μπορείς να αφαιρέσεις κάποιες λεπτομέρειες και θα πρέπει να υποβάλουμε την ε, ε, έκθεση αυτή εγκαίρως ώστε να ε, συμπεριληφθούν τα αποτελέσματα στην επόμενη πρόταση τη Κομισιόν την οποία ετοιμάζει αυτή τη στιγμή. Να μπορεί δηλαδή η Κομισιόν να λάβει υπόψη τη στη θέση του Κοινοβουλίου και αυτό θα γίνει ακόμα καλύτερα αν δεν υπάρχουν υπερβολικά πολλές λεπτομέρειες. Πάντω σα ευχαριστώ για τη συνεργασία πάνω στην έκθεση αυτή. Ευχαριστώ. Κύριος Δανέλης, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον ε, συνάδελφο Μπάχ για την καλή έκθεσή του και να επισημάνω την ε, παρότρινσή μας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει νομοθετικά μέτρα για την προστασία των επιβατών για τις συνέπειες που υφίστανται όταν μια αεροπορική εταιρεία κηρύξει πτώχευση. Ε, είναι ένα κενό και νομίζω ότι είναι σημαντικό να υπάρξει αυτή η μνήμα... Ε, γιατί μπορούμε να αναλογιστούμε ότι μονάχα μέσα στο ε, τρέχον έτος, το 2012, έχουν φτωχεύσει τουλάχιστον 7 αεροπορικές εταιρείες στην Ευρώπη. Ε, και επισημαίνω την ορθότητα αυτής μας της παρότρινσης που έρχεται σαν ένα επιπλέον ζήτημα προσκάλυψη. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Ευχαριστώ. Κύριος Κόχ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον Τζορς Μπαχ και να τον συγχαρώ. Είναι εξαιρετική η έκθεσή του. Είναι κρίσιμη η καιρή. Κατά την άποψή μου ο κόσμος μόνο για το ευρώ συζητάει. Καιρό είναι να δείξουμε ότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ο άνθρωπος, το κέντρο και πρώτα ο άνθρωπος. Γι' αυτό είναι καλή η έκθεση ε, και φέρει ισότητα ευκαιριών και για ανθρώπους ηλικιωμένους με αναπηρίες. Ευχαριστώ πολύ Ζόρος για αυτή την έκθεση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Καραμίτσος. Αλλά πριν σας δώσω το λόγο, ε, να πω και εγώ δύο λόγια. Υποστηρίζω την έκκληση του κυρίου Μπράντμπορν και άλλων. Δεν έχουμε όλοι σελίδες, ούτε είμαστε όλοι ε, κομπιουτεράδες και τρελοί με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ε, Είμαστε και παλιωμοδίτε μερικοί και χρησιμοποιούμε και ακόμα ταξιδιωτικούς πράκτορες, ταξιδιωτικά γραφεία και τέτοια. Γιατί μα ενδιαφέρουν και οι θέσεις εργασίας, όχι όλα με οθόνε. Και θα πρέπει ε, και αυτό να το έχουμε πάντα υπόψη μας. Έχω μερικές ερωτήσεις σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρώτον, έχουμε κάποια ένδειξη την οποιαδήποτε και το πότε το ΔΕΚ το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων θα αποφαθεί ε, για την προσφυγή Στέρζον. Ξέρω ότι έχει πει ο Γενικός Εισαγγελέας, αλλά οι αεροπορικές εταιρείες ε, σκεμμένα ε, καθυστερούν οποιαδήποτε πληρωμή για αποζημίωση στο Ηνωμένο Βασίλειο γιατί περιμένουν την απόφαση του δικαστηρίου. Ξέρω ότι τα δικαστήρια έχουν το δικό τους χρόνο, που δεν είναι τρένο υψηλής ταχύτητας, δεν θα το χαρακτηρίζαμε έτσι. Ε, μάλλον ο Μουτζούρης είναι ή κάποιο παλιό ε, χαλασμένο τρένο εμπορευμάτων αλλά θα είχατε καμιά χρονική έτσι, εκτίμηση. Και κάτι άλλο για το 261 για τις αερομεταφορές. Δεν ξέρω τι φρονεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά θα πρέπει να κλείσετε όλα τα παραθυράκια σχετικά με την ανωτέρα βία, διότι οι αερομεταφορές πολλές φορές κάνουν καταχρήσεις και επικαλούνται την ανωτέρα βία για να μην αποζημιώνουν τον κόσμο ως όφυλαν. 26 ώρες εγώ ε, και θα σας πω και την εταιρεία Monarch ε, είχα πρόσφατα, δεν με νοιάζει για την αποζημίωση, αλλά μου είπαν ήταν ανωτέρα βία, ε, γιατί ήταν τεχνικό και τι γίνεται με την υπόθεση στέρηση; Α, περιμένουμε, λέει, το δικαστήριο να αποφαθεί. Και ένα άλλο πράγμα που επίσης κάνει αυτή η εταιρεία, η Monarch, είναι πολύ πονηρή ε, στον τρόπο με τον οποίο υπολογίζουν το υπέρβαρο στις αποσκευές πώς να το πω, εγώ ανησυχώ έτσι και κοινωνικά και θα έλεγα ότι θα ήταν πολύ καλύτερο η γυναίκα μου και εγώ να έχουμε μία βαλίτσα και οι δυο μας, αντί δύο βαλίτσες ο καθένας στη δικιά του. Αλλά επειδή όμως η μία βαλίτσα ήταν 23 παρακαλώ κιλά, μου έφεραν το λογαριασμό 25 στερλίνες για να βάλω τη βαλίτσα μου ε, στο διάδρομο. Εγώ αντέδρασα και με παρέπεψαν στην ιστοσελίδα. Πάλι σε στέλνουν στις ιστοσελίδες. Στη σελίδα 985 κάτω-κάτω λέει ότι είναι ατομικές οι βαλίτσες. Και όχι δεν είναι ατομικές, δεν είναι ένα, ένα άτομο 20 κιλά, είναι ένα βαλίτσα. Εν πάση περιπτώσει, ε, από τον Αύγουστο ε, έχω αυτό το πρόβλημα και τα μαζεύω. Άλλο που ήθελα να αναφέρω, τα δικαιώματα των επιβατών και η πληροφόρησή τους σχετικά. Φέτος το καλοκαίρι, κύριε Καραμίτσο, έκανα σεμινάρια σε αεροδρόμια, έτσι το πέρασα το καλοκαίρι μου, και έλεγα στον κόσμο τα δικαιώματά του. Όταν είχε καθυστέρηση το αεροπλάνο. Και Brussels Airlines ήταν και μου φέραν και την αστυνομία και στη νότια Τενερίφη με τη Μόναρκ, με τη Βαλίτσα. Πολύ λίγοι από τους επιβάτες αυτούς ε, είχαν την παραμικρή ιδέα για τον κανονισμό 261. Και όταν προσπαθεί κανείς να δει την αφίσα στο αεροδρόμιο, είναι πίσω από καμιά αυτόματη μηχανή ε, που πουλάει, ή δίπλα στην τουαλέτα και κανείς δεν τη βλέπει. Μόνο σε ένα αεροδρόμιο στην Νάπολη είδα την αφίσα σε ένα σημείο ε, και μάλιστα στην οθόνη της τηλεόρασης ε, ε, στο check-in. Λοιπόν, νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε πιο πιεστικοί στον τρόπο με τον οποίο ενημερώνουμε τους επιβάτες και το ίδιο ισχύει και για τους επιβάτες των σιδηροδρόμων και άλλων μέσων μεταφοράς θα πρέπει να είναι σε εξέχουσα θέση και σε περίοπτη και όχι κάπου κρυμμένη. Και μια περίοπτη θέση, αν μου επιτρέπετε, είναι στις καντίνες ή ε, στα κυλικέ, στα εντευκτήρια εκείνων ε, που κάνουν το check-in ε, των υπαλλήλων, γιατί και αυτοί δεν έχουν ιδέα για τον οργανισμό 261. Δεν υποτίθεται ότι πρέπει να είναι μορφωμένοι, εκπαιδευμένοι, επιμορφωμένοι, καταρτισμένοι, δεν ξέρω πώς το λέτε, για να τα ξέρουν αυτοί που κάνουν το check-in και ε, την ε, εξυπηρέτηση εδάφους, ο κόσμος που δουλεύει, οι υπάλληλοι εκεί και να ενημερώνουν τον κόσμο γιατί είναι φαιά ζώνη έτσι ε, τα πάντα σε ένα αεροδρόμιο. Δηλαδή εμείς ξέρουμε τα δικαιώματά μας και οι αεροπορικές εταιρείες κάνουν ό,τι μπορούν για να ε, μην ενημερώνουν τον κόσμο. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να σταματήσουμε αυτό το παιχνιδάκι. Και συγγνώμη που επιτίθεμαι στις αεροπορικές εταιρείες, αλλά ε, πραγματικά τους αξίζει. Δεν εννοώ αυτές που εννοούσε ο Ματιό Εγκρός, αλλά το καλοκαίρι είχα σοβαρά προγράμματα με τη Monarch και αυτό συνεχίζεται. Αυτά, τα ολίγα. Ε, ποιος ήθελε το λόγο. Σύντομα, παρακαλώ. Ναι, σαν και σένα θα τα πω σύντομα. Α, συγγνώμη, εκεί. Όταν μετρήσουμε το χρόνο που αναλογεί στην κάθε πολιτική ομάδα, ε, να θυμηθούμε και κάποιον άλλο συνάδελφο που έχει δικαίωμα. Α, τον κύριο Λίχτεμπεργκ δηλαδή, εσένα. Ε, καθυστέρησε σε μια άλλη επιτροπή. Ε, άκουσα όμως την πολύ σύντομη και λακωνική σου παρουσίαση. Και μετά από αυτά θα έλεγα ευχαριστώ στον κύριο που, τον Μπαχ ε, που συμφώνησε με όλες τις ε, προτάσεις που έκανα ως ο ηγητής των Πρασίνων και ιδίως ακριβώς αυτό που ανέφερες πρόεδρε. Ότι θα πρέπει δηλαδή να έχουμε πληροφορίες σε κεντρικό σημείο, σε ένα σημείο που να είναι ορατό σε όλους και ευχαριστώ κύριε Μπακ ε, νομίζω δεν είχαμε αρκετό χρόνο στην όλη διαδικασία για να έτσι, αναπτύξουμε τις ιδέες μας. Χρειαζόταν περισσότερος χρόνος, κάτι γνώμη μου. Πάντως συγχαρητήρια, γιατί έλαβες υπόψη τις περισσότερες προτάσεις και ιδέες και ευχαριστώ που υποστήριξες και τις υπόλοιπες προτάσεις. Ευχαριστώ, Κίθ. Ο κύριος Καραμίτσος. Uh, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τις πολλές προτάσεις που διατυπώσατε. Ευχαριστώ για τις τροπολογίες των μελών της Επιτροπής. Θα πρέπει να συγχαρούμε και εμείς τον κύριο Μπακ για το έγγραφο, για τα επικοδομητικά στοιχεία που εμπεριέχει. Λίγα σχόλια ο πλευράς μου. Καταρχάς, μας ζητάτε έναν οριζόντιο κανονισμό για όλα τα μέσα μεταφοράς και οι τροπολογίες στην παράγραφο 3 είναι ευπρόσδεκτες. Συμφωνούμε απόλυτα με αυτή την ιδέα. Ε, θεωρούμε ότι τα δικαιώματα των επιβατών είναι μια ε, διαδικασία εν εξελίξη. Ε, διαφορά ανάμεσα στους τρόπους μεταφορών και στον κώδικα και τη θαλάσσια νομοθεσία που δεν έχει ακόμα τεθεί σε ισχύ ε, τι σημαίνει, ότι η πρόοδο θα γίνει σταδιακά. Δεν μπορώ να σα υποσχεθώ ότι αύριο θα έχουμε ένα κανονισμό που θα τα καλύπτει όλα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Θα διδασκόμαστε καθοδόν και βράχο πρόθεσμα μπορούμε να βάλουμε αυτό το στόχο. Η έκθεση είναι πολύ επίκαιρη, γιατί είμαστε ακριβώς σε αυτή τη διαδικασία, ψάχνουμε να βρούμε τι σημεία πρέπει να τροποποιήσουμε στην ε, νομοθεσία και ποια σημεία πρέπει να προωθήσουμε. Καταρχάς για την πληροφορία τις πληροφορίες καλύτερα. Όλοι μπορούμε να συμφωνήσουμε νομίζω ότι οι επιβάτες πραγματικά πρέπει να είναι πιο ενημερωμένοι για τα δικαιώματά τους και πώς εφαρμόζονται, πού εφαρμόζονται. Ε, πρέπει να σημειώσουμε ότι όχι όλοι μας βέβαια, αλλά κυρίως εμείς οι ασπρομάλιδες δεν είμαστε πολύ ικανοί και σαΐνια με, τα, με τις νέες τεχνολογίες, με τα iPhone κτλ. Επομένως θα πρέπει να υπάρχουν και πιο κλασικά μέσα ενημέρωσης θα πρέπει να είναι σε ευδιάκριτο σημείο, ακόμα και εκεί που ξεκουράζονται οι υπάλληλοι των ε, αεροπορίων, των αεροπο... αεροδρομίων, συγγνώμη, που ξε... Και εκεί, σε εκείνα τα σημεία, για να τα μαθαίνουν και αυτοί. Ο αντιπρόεδρος Κάλλος ε, μίλησε για αυτές τις αλλαγές στα iPhone που θα επιτρέπει να αναγράφονται οι πληροφορίες σε όλες τι επίσημε γλώσσες τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εφαρμογή αυτή, το app αυτό, ε, είναι πολύ μεγάλη ε, επιτυχία. Έχουμε ήδη ε, τέτοια ετή... Είχαμε του τελευταίους δύο μήνες 60.000 downloading αυτών των πληροφοριών. Επίσης, η εκστρατεία για τα δικαιώματα των επιβατών που είναι να εξελίξει θα παραταθεί μέχρι τέλος 2012, αρχές 2013 και επιπλέον τα 10 πιο σημαντικά δικαιώματα των επιβατών μπορεί να τα μοιράσουμε σε όλους, ούτως ώστε να αρχίσουν να μαθαίνουν α, οι επιβάτες τα δικαιώματά τους, γιατί πραγματικά υπάρχει ένα έλλειμμα ε, πληροφοριών εδώ, ο κόσμος δεν ξέρει τα δικαιώματά του, ακόμα και εγώ ο ίδιος. Κάτι μου ξεφεύγει πάντα. απλότητα λοιπόν πρέπει να το μότο μας. Πιστεύω ότι μπορούμε να σκεφτούμε και άλλα πράγματα όμως. Όχι μόνο να δημοσιεύουμε τις, τα δικαιώματα αυτά σε εύκρινα σημείο. Κοιτάξαμε κάποιες από τις τροπολογίες και πνευστήκαμε και είπαμε, αν δεν πληρώσεις... Ή μάλλον, ποτέ δεν πρέπει να είσαι σε θέση να πληρώσεις ε, στο ίντερνετ πριν κάνεις κλικ σε όλα τα άλλα σημεία τα οποία σου γράφουν ποια είναι τα δικαιώματά σου. Θα δούμε λοιπόν όλα αυτά τα σημεία πώς μπορούμε να τα βελτιώσουμε, τις πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τις υποχρεώσεις που έχουν οι αερομεταφορικές εταιρείες για να δίδουν ε, σαφείς πληροφορίες. Ε, αυτό σημαίνει περισσότερος διάλογος μεταξύ των επιβατών και των ε, μεταφορικών εταιρεών. Φυσικά, μην ξεχνάμε ότι ο φτωχό, επιβάτης, ο κακομύρης, ο επιβάτης που εμφανίζεται μπροστά στο, στον κισέ εκεί του υπαλλήλου, κάλλιστα μπορεί να είναι σε μειονεκτική θέση σε σχέση απέναντι στον υπάλληλο. Αλλά πρέπει να είναι ακριβείς οι πληροφορίες και όχι παραπλανητικές. Πάμε τώρα στη διαφάνεια. Υπάρχουν πολλές τροπολογίες Παράγραφος 11 για την ε, διαφάνεια των τιμών. Χαιρόμαστε για τις πολλές αυτές τροπολογίες. 13 βουλευτές έκαναν προτάσεις για αυτό το σημείο. Αυτό δείχνει ότι είναι μια μεγάλη ανησυχία για πολλούς πολίτες. Εδώ πρέπει να και να μάθουμε και να διδαχτούμε. Τώρα ε, τσεκάρουμε τη σχετική νομοθεσία για να δούμε αν είναι κατάλληλη και αν πρέπει να τροποποιηθεί. Κοιτάμε λοιπόν αυτές τις τροπολογίες. Πάντως η διαφάνεια είναι ένα θέμα το οποίο παρακολουθούμε εκ του σύνεγγης. Σε αυτά τα πλαίσια της προσπάθειας ελέγχου της καταλληλότητας της νομοθεσίας. Και θα επανέλθουμε εν ευθέτω χρόνο. Για την ε, εφαρμογή. Το άλλο θέμα που θέτει η έκθεση. Βεβαίω θα πρέπει να εφαρμοστούν σωστά τα δικαιώματα, το λέει η έκθεση, αλλιώ έχουν νόημα. Συμφωνούμε απόλυτα με αυτό. Φυσικά, ε, σήμερα οι επιβάτες μπορούν να παίρνουν πληροφορίες τα δικαιώματά τους από τις εθνικές αρχές ε, και μπορούν να ζητήσουν περαιτέρω βοήθεια, μπορούν να πάρουν πληροφορίες χωρίς περαιτέρω κόστος μέσα, μέσω διαφόρων οδών. Παραδείγματος χάρη υπάρχει ένα κέντρο άμεσης επαφής με ένα δωρεάν νούμερο που δίνει πληροφορίες σε όλες τις επίσημες γλώσσες μας. θα πρέπει να αναφέρουμε και το δίκτυο ECC και αυτό το κέντρο άμεσης έτσι, πληροφορίας, πληροφόρησης. Γιατί όντω πρέπει να καταρτήσουμε κάποιου ανθρώπου για να εκπαιδεύσουμε κάποιου ανθρώπου για να δίνουν αυτέ τι πληροφορίε. Επίση, ε, ο χειρισμό παραπώνων ε, και η τροποποίηση του κανονισμού 261. Σας ευχαριστούμε την προσοχή στη μελλοντική νομοθεσία για την επίλυση των διαφορών ε, στο διαδίκτυο και τον εναλλακτικό τρόπο επίλυσης διαφορών. Ε, γιατί χάρη και στις αρχές ε, στο ECC, σε αυτό το κέντρο, αλλά και σε αυτούς τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης διαφορών θα λυθούν πολλές υποθέσεις. Άλλα θέματα που θέσατε είναι η δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού εντύπου για όλα τα, τους τρόπους μεταφορών, για παράπονα που μπορεί να υπάρχουν κτλ. Θα το επεκτείνουμε σε όλους τους τρόπους ε, αυτό που έχουμε. Υπάρχουν και άλλες ε, τροπολογίες πολύ σημαντικές που συνδέονται με, με την πολιτική no-show, δηλαδή τι θα γίνει τον επιβάτη αν δεν εμφανιστεί. Δηλαδή, ε, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το εισιτήριο επιστροφή αν δεν έχει πάει, α πούμε. Πρέπει να δούμε ε, πώ ε, θα περιορίζουμε τι ε, αεροπορικέ εταιρείε να μην κάνουν καταχρήσει όταν χρησιμοποιούν τέτοιε πολιτικέ. Τώρα, οι ευθύνε. Ο κανονισμός 261 έχει πρόβλημα εδώ διαφάνειας για τα δικαιώματα. Εδώ θα το αναγνωρίζουμε. Θα πρέπει να ενισχύσουμε και την εφαρμογή ω προ αυτό. Και σε αυτή τη ε, μεταρρύθμιση του κανονισμού θα διευκρινίσουμε και τα δικαιώματα των ε, επιβατών, αλλά και την έννοια των έκτακτων συνθήκων που πολύ αναφέρατε. Πρέπει να το ψάξουμε αυτό το θέμα και να προσπαθήσουμε να δούμε πώς αντιμετωπίζετε, να αντιμετωπίζετε με διαφανή τρόπο, ούτως ώστε να μην χρησιμοποιείτε ως δικαιολογία για να μην αποζημιώνουν τους επιβάτες οι αεροπορικές εταιρείες, οι γενικά. Η νομοθετική όμως πρόταση δεν νομίζω ότι θα μας επιτρέψει ε, ένα θέτο χρόνο να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Έχουμε τον 261 και τον 1008. Ε, ε, γι' αυτό χρειάζονται, χρειάζεται σωστή εφαρμογή αυτών των κειμένων και για να εφαρμοστούν σωστά το Κοιτάμε τώρα να δούμε λύσεις για τους ε, επιβάτες που μπορούν να εφαρμοστούν αποτελεσματικά στο εγγύς μέλλον. Γι' αυτό μέχρι το τέλος του 2012 θα κάνουμε κάποιες ε, προτάσεις το πολύ πολύ αρχές του 2013. Κάποια άλλα σημεία που αναφέρθηκαν. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα βγάλει την απόφαση του πριν από το τέλος του 2012, ελπίζουμε, αναφέρθηκα στην ε, ανωτέρα βία. Πολύ συχνά το χρησιμοποιούν για, ως παραθυράκι διαφυγής. Εγώ δεν ήξερα. Αυτό που αναφέρατε εσείς, Πρόεδρε, για τα 23 κιλά σε μία βαλίτσα. Πολλοί είναι πανέξυπνοι έτσι και προσπαθούν να βρουν τρόπους να γλιτώσουν τις υποχρεώσεις τους, όντως. Ο κύριος Τέιλον ανέφερε την ανάγκη να υπάρχουν πληροφορίες ευκρινέ σημείο. Πρέπει τέλος πάντων να υποχρεώσουμε τις ε, εταιρείε να εφαρμόζονται να, εφαρμόζουν τα δικαιώματα των επιβατών. Το 4α, το 6, 21, 9, όλες αυτές τις τροπολογίες είναι βελτιωτικές ως προς το κείμενο, τις υποστηρίζουμε. Η έκθεση και οι τροπολογίε ήταν πολύ χρήσιμε για μα, ακριβώ γι' αυτό. Ο βασικό στόχο είναι τα δικαιώματα των επιβατών να είναι κατανοητά, είναι σημαντικέ οι πληροφορίε γι' αυτό και θα πρέπει να ενισχυθεί η εφαρμογή του σε όλου του τρόπου μεταφορών, τόσο ώστε να υπάρχει μια συγκλίνουσα προσέγγιση σε αυτόν τον τομέα. Η Κομισιόν θα συνεχίσει την δουλειά της για τα ρυθμιστικά και μη ρυθμιστικά θέματα, ούτως ώστε να ενισχύσει την, ε, τα δικαιώματα, ούτως ώστε ε, η νομοθεσία να εφαρμόζεται με αποτελεσματικό τρόπο ε, και αναλογικό, να λαμβάνουμε υπόψη μας επιβάτες με δικές ανάγκες, άτομα. Και θα λαμβάνουμε υπόψη μας και τις στατιστικές, ούτως ώστε να δούμε πού χρειάζεται δράση. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Μπάχα, έχετε τίποτα να προσθέσετε. Πολύ σύντομα, διότι ο χρόνος περνάει. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για τους επένους και την υποστήριξή σας. Ε, όσον αφορά τις παρατηρήσεις της Κομισιόν, ανέφερε αναλυτικά, ε, αναφέρθηκε αναλυτικά στο θέμα αυτό και αποδεικνύει έτσι ότι παίρνει στα σοβαρά το θέμα αυτό και ε, πρόκειται να υποβάλει ενδιαφέρουσες προτάσεις στο εγγύς μέλλον. Ε, συμφωνώ με τους ε, διάφορους βουλευτές που ζητάνε σαφήνεια, επιπλέον πληροφορίες και θα ήθελα στη συνάδελφο Σαρισάρ και σε άλλους ε, να πω ότι δεν έχω πρόβλημα με τους ε, πιο ηλικιωμένους ε, και αυτό που λέμε για τα smartphone applications, ε, για τις εφαρμογές για τα προηγμένα τηλέφωνα. Θα πρέπει οι πληροφορίες να παρέχονται στην γλώσσα του καταναλωτή, επίσης στα άτομα με περιορισμένη κινητικότητα. Πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε σαφείς κανόνες. Σαφείς κανόνες θα πρέπει να έχουμε, όπως και τις εύλογες προσαρμογές και ε, πρόσφατα έστειλα μια επιστολή στον ε, Επίτροπο Κάλλας όσον αφορά ε, τα μουσικά όργανα στα αεροπλάνα. Θα πρέπει να υπάρχει σαφήνεια για τους επιβάτες. Σας ευχαριστώ για την υποστήριξή σας. Ευχαριστώ, Ζορς. Ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί αύριο. Όπως σας είπα, θα πρέπει να φροντίσουμε να ε, φτάσει το θέμα στην ε, ημερήσια διάταξη της Ολομέλειας. Ε, γι' αυτό επαναλαμβάνω την εκκλησή μου. Το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξή μας είναι ο Επίτροπος Σιμ Κάλασε για, τις, για τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων. Έχουμε 45 λεπτά μόνο διότι πρέπει να προλάβει αεροπλάνο. Ελπίζω να μην είναι βρετανική πτήση διότι τότε σε περίπτωση καθυστέρησης δεν θα λάβεις αποζημίωση όσον αφορά λοιπόν την οδηγία για ε, τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων. Παρακαλώ. Ε, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί βουλευτές, ε, σας ευχαριστώ και πάλι για τη δυνατότητα αυτή να έχουμε σήμερα ανταλλαγή απόψεων σχετικά με ένα πολύ σημαντικό θέμα. Στο Βερολίνο θα πάω να, να μιλήσω για τους σιδηρόδρομους. Mm. Γιατί μιλάτε, γιατί γελάτε. πρόταση σχετικά με τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων. Ε, σήμερα θα πεθάνουν πέντε άνθρωποι στους δρόμους ε, της Ευρώπης ως αποτέλεσμα ατυχημάτων που σχετίζονται με τεχνικά προβλήματα. Ε, το 6% των σοβαρών ατυχημάτων των αυτοκινήτων οφείλονται σε τεχνικά προβλήματα και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στόχο να μειώσει στο μισό τα ε, ατυχήματα στους δρόμους μέχρι το 2020 και να ε, πέσουν στο 0 το 2050. Ε, βλέπουμε ότι έχει επιβραδυνθεί η ότι, ότι έχουν μειωθεί οι θάνατοι στους δρόμους. θα πρέπει όμως να καταβάλουμε προσπάθειες για να πετύχουμε τους στόχους μας μέχρι το 2020. Το να ε, πηγαίνει κανεί το αυτοκίνητο του στο δεν, είναι, δεν γίνεται για λόγου. λόγους. Ε, σώζει ζωέ αυτό ο τεχνικό έλεγχο. Εάν οδηγάτε όχημα το οποίο ε, δεν είναι κατάλληλο για οδήγηση στου δρόμου, τότε αποτελείται κίνδυνο για τον εαυτό σας και για οποιονδήποτε άλλο βρίσκεται στο αυτοκίνητο, την οικογένειά σας, τους φίλους σας. Κινδυνεύουν όμως και όλοι οι άλλοι χρήστε στο δρόμο γύρω σας στην Ευρώπη. Είναι πολύ απλό. Δεν θέλουμε λοιπόν ε, αυτά τα ε, δυνάμει ε, θανατηφόρα αυτοκίνητα στους δρόμους μας. Τι κάνουμε λοιπόν, έχουμε περιοδικούς τεχνικούς ελέγχους, έχουμε τεχνικούς ελέγχους των εμπορικών οχημάτων και τροποποίηση της οδηγίας για τους τεχνικούς ελέγχους. Τα δύο πιο σημαντικά νομοθετήματα θα γίνουν κανονισμοί για να έχουμε καλύτερα, καλύτερο επίπεδο πρότυπων ελέγχων για, ως βάση για την μελλοντική αμοιβή αναγνώριση. Τρία βασικά ε, στοιχεία έχουν να κάνουν με τους ε, περιοδικούς τεχνικούς ελέγχους. Ε, πρώτον, θέτουμε νέα ελάχιστα πρότυπα σχετικά με την ποιότητα των ελέγχων και των ελεγκτών. Όταν πληρώνετε 40 ευρώ για τον έλεγχο στο κταίο, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν παίρνετε απλό ένα πιστοποιητικό, αλλά γίνεται και σωστός και υψηλής ποιότητας έλεγχος στο όχημά σας. Αυξάνουμε την συχνότητα των ελέγχων για τα παλαιά αυτοκίνητα ή αυτά ε, που έχουν ε, κάνει πολλά χιλιόμετρα. Τα ε, σημερινά αυτοκίνητα γίνονται όλο και πιο ασφαλή, αλλά τα παλαιότερα αυτοκίνητα άνω των 6 ετών συνδέονται με περισσότερα ατυχήματα και πιο σοβαρά ατυχήματα. Για ε, τα ε, ε, επιβατικά αυτοκίνητα, ο πρώτος έλεγχος θα πρέπει να γίνεται μετά από τέσσερα χρόνια, ο δεύτερος μετά από δύο χρόνια και μετά κάθε χρόνο. Αυτό θα αντικαταστήσει τους παρόντες κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαιτούν έλεγχο κάθε δύο χρόνια μετά την εξαετία. Ωστόσο, τα περισσότερα κράτη-μέλη απαιτούν ήδη ετήσιο έλεγχο πολλών οχημάτων. Τέλος, έχουμε υποχρεωτικό έλεγχο για μοτοσυκλέτες και μοτοποδήλατα. Οι μοτοσυκλετιστές ε, είναι ε, ομάδα, ε, με, ομάδα υψηλού κινδύνου, σχετίζονται με πολλούς θανάτους, πάνω από 2.500 άτομα σκοτώνονται κάθε χρόνο. Γύρω το, Περίπου το 8% των αχημάτων όπου εμπλέκονται μοτοσυκλέτες έχουν να κάνουν με τεχνικά προβλήματα αν εφαρμόσουμε ελέγχους σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση θα σώσουμε 270 ε, ζωές ε, και ε, θα αποφεύγουμε 3.000 σοβαρούς τραυματισμούς το χρόνο. Θα ήθελα επίσης να αδράξω την ευκαιρία να ξεκαθαρίσω το θέμα των ιστορικών οχημάτων. Δεν έχουν κανένα λόγο να ε, φοβούνται το, την πρότασή μας. Ε, ο ορισμός που χρησιμοποιούμε βασίζεται ε, στην χρήση των ανταλλακτικών, τα ιστορικά ε, στοιχεία και την ανάγκη να μην αλλάζουν τα ιστορικά χαρακτηριστικά των βασικών ε, στοιχείων του αυτοκινήτου όπως είναι η μηχανή και τα φρένα για να διατηρηθεί η ιστορική αξία των οχημάτων αυτών. Ε, Παρ' όλα αυτά ε, είναι δυνατόν να τροποποιηθούν τα αυτοκίνητα ή να χρησιμοποιηθούν μη, βασι... μη, μη ε, πρωτότυπα ε, ανταλλακτικά εφόσον μπορεί κανείς παρόλα αυτά να πετύχει έγκριση. οι ε, ιδιοκτήτε παλαιών αυτοκινήτων δεν σημαίνει αυτό ότι δεν μπορούν να ε, κάνουν τροποποίηση στα αυτοκίνητα του. Ε, ωστόσο, αν επιλέξουν να βάλουν σύγχρονη μηχανή σε ένα αυτοκίνητο του 1950 ε, με μεγαλύτερη ισχύ, τότε η Κομισιόν θεωρεί ότι η ασφάλεια ενός τέτοιου αυτοκινήτου θα πρέπει να διασφαλίζεται με τακτικούς ελέγχους. Ε, κατά τους ε, επιτόπου ελέγχους, τους ελέγχους στο δρόμο των αυτοκινήτων υπάρχει άλλο ένα στοιχείο. Θέλουμε να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα αυτών των ελέγχων. προτείνονται νέα ελάχιστα πρότυπα για τους ελέγχου, για τους ελέγχους αυτούς και θα πρέπει να γίνονται στοχευμένοι έλεγχοι ε, εταιριών ε, με ε, κακό ιστορικό όσον αφορά την ασφάλειά τους. Ελπίζω ότι η συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πάνω στη σημαντική αυτή πρόταση θα μπορέσει να ξεκινήσει σύντομα και να υιοθετηθεί σύντομα η πρόταση. Θα ήθελα επίσης να σας θυμίσω ότι η πρόταση αυτή αναμένεται να σώζει πέντε ζωές στην Ευρώπη κάθε μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ ο Γκρό, Γκρός Για να απαντήσει και ο επίτροπο. έχουμε μισή ώρα. Λιγότερο από μισή ώρα. Το έχετε υπόψη σας ο κύριος Γκρός. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για την πρόταση. Νομίζω ότι πραγματικά ε, γράφεται στο πλαίσιο των όσων είχαμε εδώ επεξεργαστεί και στην αρχή και μετά στη Λευκή Βίβλο για την οδική ασφάλεια που πρέπει να είναι κέντρο βάρου στην πολιτική μας. Είναι γεγονός ότι δείχνουμε και μπορούμε να δείξουμε ότι η ευρωπαϊκή πολιτική είναι πολύ κοντά στον πολίτη. Γι' αυτό περιμένουμε από την παρούσα νομοθεσία γρήγορα βήματα, συγκεκριμένα αλλά και αποτελεσματικά. Τα τεχνικά στοιχεία είναι βεβαίω τμήμα τη οδική ασφάλεια. Απλώ θέλω να θυμίσω ότι η συζήτηση που κάναμε εδώ για τα ναρκωτικά, ε, το αλκοόλ, την ταχύτητα και τι υποδομέ στο παρελθόν οδήγησε και ε, σε περαιτέρω ε, συζήτηση. Βεβαίως ο τεχνικό έλεγχο είναι σημαντικό. Για τα διασυνοριακά και να μας συμπεφάτε θα μιλήσω εγώ, δεν σα εκπλήσει. Για μένα είναι πολύ σημαντικό να έχει την ίδια ποιότητα σε όλες τις χώρες ο τεχνικός έλεγχος, αλλά και η κατάρτιση των επιθεωρητών και των ελεγκτών. Και επίσης διασυνοριακά να μπορεί κανείς να ελέγχει την ποιότητα αυτή. Ένα απλό παράδειγμα να σας δώσω φορτηγά από μακρινές χώρες ξαφνικά έρχονται στο κτέο το Σαββατοκύριακο που δεν μπορούν να φύγουν και να ξανάρθουν. Πώς κάνουμε τον έλεγχο των ελεγκτών εμείς. Αλλιώς είναι ένα κομμάτι χαρτί που δεν αποδεικνύει τίποτα. Υπάρχουν καλά παραδείγματα από το μικρό μας Βέλγιο ε, που έχουμε ε, εισαγάγει ε, ένα καρπάς ένα, ε, σύμβαση ας πούμε ε, μεταξύ ε, ενός παρόχου υπηρεσιών και του οδηγού για να είμαστε βέβαιοι ότι είναι πάρα πολύ σωστές οι ενδείξεις που αναγράφονται σε αγοραπολισίες αυτοκινήτων. Προσπαθώ να τραβήξω την προσοχή των φιλελευθέρων, γιατί δεν έχουν γράψει κανένα να μιλήσει. Ο κύριος Αλχαντράουι, για δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον Επίτροπο για την εισαγωγή. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό και το βλέπω ότι του δίνει και τη δέουσα προσοχή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με την ησυχία μας θα τα μελετήσουμε, θα τα συζητήσουμε αυτά. Είναι προφανές και δεν χωράει καμία αμφιβολία ότι η οδική ασφάλεια ε, μπορεί να επιτευχθεί και από μεγαλύτερη τυποποίηση και ε, μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε σε αυτά. Επίσης συμφωνούμε ότι πρέπει να αυξηθεί ο ρυθμός των τεχνικών ελέγχων και η συχνότητα, αλλά και η ποιότητά τους να εναρμονιστεί. Γνωρίζουμε όλοι ότι υπάρχουν κράτη-μέλη που, ε, να παίρνουν τα πράγματα πιο σοβαρά από κάποια άλλα και είναι σημαντικό να μπει λίγο πιο ψηλά ο πύχης με τη βαρούσα νομοθεσία. Και χαίρομαι για αυτά που λέτε για τα δίκυκλα, τα μοτοποδήλατα και τις μοτοσικλέτες. Μας αναφέρατε και τον αριθμό των νεκρών και των ε, τραυματίων. Ε, λίγο για τις εταιρείε που έχουν κακή φήμη ε, και θα πρέπει να ελέγχονται. Εντάξει, αυτό είναι καλή αρχή, αλλά είναι πολύ σημαντικό επίσης να δούμε ποιος είναι ο ορισμός. Τι εστί καλή εταιρεία, κακή εταιρεία. εταιρεία. Θα πρέπει να εναρμονιστεί λίγο και ο ορισμός και ο χαρακτηρισμός. Έτσι ώστε να μην έχουμε κάποια κράτη-μέλη που να συγκεντρώνουν πάρα πολλές εταιρείε που χαρακτηρίζονται κακές ενώ κάποια άλλα κράτη-μέλη να έχουν μόνο καλέ εταιρείε όταν δεν ανταποκρίνεται αυτό στην πραγματικότητα. Αυτά, μερικέ μόνο παρατηρήσει. Σταματώ εδώ, αλλά πιστεύω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε και σε γενικέ γραμμέ συμφωνούμε. Ο κύριο Ντεμπάκερ από του Φιλελευθέρου για δύο λεπτά. Ξυπνήσαμε, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Επίτροπε, και εμεί σα ευχαριστούμε για τι προτάσει σα, για τι εξηγήσει σα. Ε, μα φαίνεται πολύ σημαντική και εμά η πρόταση αυτή για να μπορέσει όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει τις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές και την ασφάλεια. Γιατί θα πρέπει να προσέχουμε καλύτερα τα οχήματά μας. Δύο-τρία ε, σύντομα. Εκτός από τους ισχυρούς ελέγχους στα ΙΟΤΑΧΗ, θα πρέπει να έχουμε ισχυρούς και καλύτερους ελέγχους στα δίκυκλα και τρίκυκλα. Εμείς ως φιλελεύθεροι φοβούμαστε με αυτά που προτείνετε, γιατί μπορεί να είναι πολύ καλή η ιδέα σας για να ε, πριτανεύει και εκεί η ασφάλεια, αλλά θα πρέπει οπωσδήποτε να δούμε τι γίνεται και με το διοικητικό φόρτο και τη γραφειοκρατία. Ε, θα πρέπει να παραμείνουμε προσγειωμένοι και ρεαλιστές. όχι μόνο τα τεχνικά ζητήματα να σκεφτόμαστε και τις ε, υποδύναμη ας πούμε, αλλά ε, υπάρχουν και άλλα θέματα ασφαλείας που είναι οι υποδομές και οι δρόμοι. Και ε, ίσως να σας αναφέρω και ένα μικρό περιστατικό αν θέλετε, για τα λεγόμενα ιστορικά αυτοκίνητα, τις αντίκες. Έχουμε πολλούς ε, που ενδιαφέρονται και οπαδούς που ασχολούνται με αυτά τα αυτοκίνητα. Γενικά σας υποστηρίζουμε και σας ευχαριστούμε που ήρθατε εδώ. Για δύο λεπτά ο κύριος Κράμερ, Μάικλ. Βεβαίως είναι σημαντική ε, η υπόθεση. Κάθε χρόνο έχουμε 70.000 νεκρούς. Η καταστροφή του τσουνάμι που ήταν, ε, η καταστροφή του αιώνα ήταν 200.000. Ε, ε, στην Ευρώπη που έχουμε 500.000 νεκρούς το χρόνο, καταλαβαίνετε, ε, συγγνώμη, 50.000 έχουμε ένα τσουνάμι κάθε 4 χρόνια. Ε, Βεβαίω τα πιο καινούργια αυτοκίνητα να μην τα ελέγχουμε τόσο συχνά, τα πιο παλιά ναι. Ε, θα ήθελα στοιχεία, τι γίνεται σε κάθε χώρα ε, αναδιετία κάθε χρόνο που υπάρχει αυτή η κατάσταση για να μπορέσουμε να κάνουμε και τις συζητήσεις και να εξηγούμε στις χώρες μας τι γίνεται. Και σας παρακαλώ. Κάτι θέλω να επικρίνω όμως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κύριε Επίτροπε, θα θυμάστε ίσως σας είχαμε δώσει ένα ωραίο φυλάδιο. Πριν από 25 χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, αγωνιζόταν για περιορισμό του ορίου ταχύτητας. Γιατί ε, είναι η μεγαλύτερη κίνδυνη στην Ευρώπη. Σας δώσαμε ένα φιλαδιάκι αλλά την τελευταία 25 ετία δεν έκανε τίποτα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επανειλημμένα το φέραμε. 110, 120, 130 είναι το όριο ταχύτητας στους αυτοκινητοδρόμους. Στη Γερμανία δεν υπάρχει κανένα όριο απολύτω και εδώ χρειάζεται συντονισμός και ευρωπαϊκός και στις πόλεις που έχουμε 50 ε, χιλιόμετρα όριο ταχύτητας. Οι περισσότερες ε, πόλεις όμως έχουν σήμερα όριο στους δρόμους τα 30 χιλιόμετρα. Παρακαλώ όχι μόνο τα τεχνικά τεχνικά στοιχεία που έχουν σημασία, αλλά να έχουμε υπόψη μα και τα άλλα. Δεν χρειαζόμαστε μόνο έξυπνα αυτοκίνητα, χρειαζόμαστε και έξυπνου οδηγού, που καμιά φορά είναι τόσο ηλίθιοι που πατάνε του ποδηλάτε. Η κυρία Φώστερ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ την Κομισιόν που ήρθε εδώ για να μιλήσει για αυτό το πακέτο. Είναι η κατάλληλη στιγμή για να μιλήσει γι' αυτό. Ένα-δύο στοιχεία Φυσικά υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες για τους ελέγχους. Είναι πολύ σωστό ότι θα πρέπει να έχουμε τακτικούς ελέγχους των οχημάτων και ότι τα παλιότερα οχήματα ε, είναι αυτά που στραβούν περισσότερο. Στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε ένα κταίο κάθε τρία χρόνια. Ε, ε, κάθε τρία χρόνια, ειδικά τα οχήματα που έχουν πολλά χιλιόμετρα, ε, τα τσεκάρουμε. Κανονικά όμως ε, μετά την τριετία θα πρέπει να ελέγχονται κάθε ένα χρόνο. Ε, επίσης ε, με τους χώρους των κτέων δεν έχω κανένα πρόβλημα, οι χώρες τα ρυθμίζουν. Ε, επίσης δεν πρέπει να περιμένουμε 6 χρόνια για να ελεγχθεί για πρώτη φορά ένα όχημα. Είναι πολύ μεγάλο ε, το χρονικό διάστημα για τις αντίκες. Ε, νομίζω εντάχθηκε πολλές πιέσεις η Κομισιόν ήδη λάβαμε πάρα πολλά email και εμείς οι ευρωβουλευτές από τους οπαδούς των, του είδους αυτού. Ε, φυσικά δεν θέλουμε να αλλάξουμε αυτά τα οχήματα. Έχουμε πολλούς θειασότες τους που κάνουν πολλή δουλειά σε αυτά και για πολλούς λόγους, γιατί υπάρχει και αγορά αυτών των οχημάτων, πρέπει να διατηρηθούν αυτές οι αντίκες. Αυτό που θέλω να πω είναι το θέμα της, των ανθρώπων που ασχολούνται ίδιοι όσοι έχουν τέτοιε αντίκε ασχολούνται ίδια με τα οχήματα. Δεν θέλω λοιπόν να τους, μπλέξουμε, να τους περιπλέξουμε το βίο. Ευχαριστώ λοιπόν την Κομισιόν συνολικά για την προσπάθειά της. Ε, είναι ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Δεν θέλουμε υπερβολική νομοθεσία, υπερβολικούς ελέγχους όταν δεν χρειάζονται αυτοί. Θα πρέπει να είναι απλή η έλεγχη, και οι κανόνες αφή, ούτως ώστε να μην επιβάλλουμε περιττό Περιτές πάνε σε ανθρώπους. Ο κύριος Κόκ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Οι ε, εκθέσεις πρωτοβουλίας είναι χρήσιμες ε, διότι ε, στην δική μου περσινή τέτοια ζητήσαμε από την Κομισιόν να υποβάλει ένα σχετικό πακέτο. Όσον αφορά τους ε, εμπειρογνώμονες, ε, χρειαζόμαστε ελάχιστα πρότυπα, χρειαζόμαστε και ελάχιστα πρότυπα όσον αφορά τις μεθόδους ελέγχου. Ερώτηση, τα κράτη-μέλη μπορούν να προχωρήσουν πέρα από αυτές τις ελάχιστες απαιτήσει και με το πακέτο αυτό μπορούμε να κινητοποιήσουμε την έρευνα και την ανάπτυξη στην Ευρώπη ώστε τα κταίω αυτά να είναι ε, υψηλότερης ποιότητας και να πραγματοποιούνται πιο αποτελεσματικά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Τίτερ. Ο κύριος Ερτούκ. Ε, ε, λείπει κύριος παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ με τους άλλους ομιλητές. Καλωσορίζω την πρόταση της Κομισιόν. Γενικά οι προτάσεις είναι καλές. Ε, θα πρέπει να μειωθούν οι εκπομπές του άνθρακα και άλλων ρήπων. Πολύ καλό. Ε, το θέμα της απάτης που γίνεται με τα χιλιόμετρα των αυτοκινήτων έχει τεθεί. Ε, και ξέρω πολύ, πολύ καλά ότι είναι δύσκολο οι καταναλωτές να ενημερωθούν σωστά για τον αριθμό των χιλιόμετρων των ε, αυτοκινήτων δεύτερου χεριού, που πουλούνται δεύτερο χέρι. Γιατί γίνονται απάτες. Θα πρέπει αυτό το διαβατήριο των αυτοκινήτων να χρησιμοποιείται όχι μόνο στην Ιρλανδία, αλλά σε όλη την Ευρώπη. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει γενικά εμπιστοσύνη σε όλο τον κλάδο ε, και όχι απλή γραφειοκρατία. Ε, επίσης για τα φορτηγά. Ε, φοβάμαι πως αυξηθεί απλώς η γραφειοκρατία για τα φορτηγά. Για αυτό το σημείο της Κομισιόν έχω πρόβλημα. Και για τα κοινά πρότυπα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ό,τι αφορά τα κέντρα ελέγχου, είναι πολύ σημαντικό γιατί στη χώρα μου, ε, σε ένα κέντρο ελέγχου στο Δουβλίνο, ανακαλύψαμε ένα δίκτυο απάτης. Επομένως, θα πρέπει να ελέγχουμε αυτές τις εταιρείες που κάνουν τους ελέγχους. Ο κύριο Σαρτούκ τώρα, ευχαριστώ Πρόεδρε ε, και συγχαρητήρια προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρόταση αυτή που ήταν πραγματικά απαραίτητη και ιδιαίτερα ευχαριστώ που έχετε βάλει και τις μοτοσυκλέτες ε, στην πρόταση. Είναι πραγματικά σωστό αυτό προς την ορθή κατεύθυνση. Εγώ περισσότερο έχω ερωτήσεις κύριε Επίτροπε για να μπορέσω να το καταλάβω. Αναφερθήκατε στις ελάχιστες προδιαγραφές και πρότυπα. Μέχρι τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει φροντίσει να εφαρμόσει και να αναλύσει ε, τα πρότυπα που ισχύουν μέχρι τώρα. Ναι, ε, τι απορίσματα έχετε βγάλει. Δεύτερον, στο παράρτημα 6, αν δεν απατώμε, αναφέρονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τι αναμένεται. Στην εναρμόνιση ε, είναι πάντα προσαρμογή το θέμα και αυτό θα ήταν ενδιαφέρον για χώρες που έχουν υψηλά πρότυπα θα συναντηθούν πουθενά στη μέση αν συναντηθούν οι χώρες για να εναρμονιστούν για τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Ε, στη Γερμανία υπάρχουν συγκεκριμένοι ε, μηχανικοί που μπορούν να ελέγξουν, όχι όλοι. Στις άλλες χώρες τι γίνεται. Όταν γίνει κάποια αλλαγή Δηλαδή, όταν αλλάζει χέρια στη μεταβίβαση, αν έχει περάσει κταίο πριν από δύο μήνε, γιατί πρέπει στη μεταβίβαση να ξαναπεράσει κταίο, δεν το καταλαβαίνω. Επίση, για του ιδιώτε αναφέρεται ότι ενδεχομένω θα μπορούσαν να ελέγχουν ιδιωτικό κταίο. Αυτό μου φαίνεται πάρα πολύ προβληματικό. Δηλαδή, κάποιο που δεν είναι κταίο, που είναι αντιπροσωπή αυτοκινήτων, να μπορεί να εκτελεί και χρέη ελεγκτού προβληματικό μου φαίνεται. Στο άρθρο 17 λέτε ε, κάτι εξουδιώτηση πράξης. Ε, ανάλογα με την τεχνική πρόοδο και την τεχνολογία θα πρέπει να ε, αφήνεται αυτό στη διακριτική ευχέρεια. Όχι, θα πρέπει να το Εντάξει, και το κοινοβούλιο, γιατί τι θα πει η τεχνολογική πρόοδος. Και αυτή η ρύθμιση 1 στη Γερμανία αφορά 50% των ε, Ιωταχή. έχετε κάνει μελέτη αντικτύπου, εάν αυξάνεται έτσι η οδική ασφάλεια ή όχι. Για τελευταίο, το κόστος. Γιατί μετά την επταετία το να πρέπει να πηγαίνει στο αυτοκίνητό σου κάθε χρόνο στο κτέο, το θεωρώ και αυτό προβληματικό. Ευχαριστώ. Κύριος Πάκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να κάνω κάποιες θετικές παρατηρήσεις. Ε, καταρχήν, ε, Βρίσκω την πρόταση να έχουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο ελέγχους πολύ καλό διότι έτσι μπορούν να εφαρμόζονται ενιαία τα πρότυπα. Το θέμα. Ο νόμος ε, είναι πώς μπορούμε να το εφαρμόσουμε αυτό ενιαία, διότι ε, ε, επανειλημμένα υιοθετούμε τα πρότυπα, αλλά τελικά στην εφαρμογή κολλάμε και στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να αποφύγουμε το πρόβλημα αυτό. Και Επίσης, ε, τους ενιαίους αυτούς ελέγχους, ε, τα ενιαία πρότυπα βρίσκω ότι είναι προϋπόθεση για την ε, μεταφορά των οχημάτων. Και μία ερώτηση τέλος. Παρότι υπάρχουν υψηλά πρότυπα για τα οχήματα, θα μπορούσατε να φανταστείτε το πρόβλημα της ε, Μήπως θα μπορούσαμε να έχουμε ενιαίες ε, προϋποθέσεις σχετικά με τον εξοπλισμό ασφαλείας που θα πρέπει να έχει μαζί το ένα αυτοκίνητο ώστε να μην ε, ζητάει το ένα κράτος κάποια πράγματα και σε άλλο κράτος να ζητάμε άλλα πράγματα. Έτσι θα μπορούσαμε να έχουμε μια χρήσιμη απλοποίηση των κανόνων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πίρκερ. Κυρία Αγιάλα Σέντερ, δύο λεπτά. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρόταση. Παρόλο που υπάρχουν μερικά στοιχεία που μας προβληματίζουν. Τώρα που ζούμε και σε κρίση ιδιαίτερα στη χώρα μου, παλιώνουν πάρα πολύ γρήγορα τα αυτοκίνητα. Ε, δηλαδή είναι πιο παλιά τα αυτοκίνητα από οδηγεί ο κόσμος. Και ακριβώς υπάρχει πρόβλημα οδικής ασφάλειας ε, και ίσως χαλαρώνουν και τα μέτρα που λαμβάνονται και η συνειδητοποίηση του κοινού. Θα μπορούσε να μας πει ο Επίτροπος κάτι για τις χώρες που πιέζονται πιο πολύ σήμερα από την κρίση. Τι γίνεται Μήπως θα μπορούσατε να βοηθήσετε λίγο για την ε, απόσυρση ας πούμε που ε, βοηθάει τον κόσμο να αλλάξει αυτοκίνητο, να ανανεώσει το, ο στόλος των οχημάτων που κυκλοφορεί ε, και μέσω του κτέου. Ε, μια που είστε εδώ όμως κύριε Κάλλας. Θα μπορούσατε να μας πείτε λίγο και για την τεχνική αρτιότητα των αεροσκαφών, γιατί με τη Ryanair έχουμε πρόβλημα στην Ισπανία και θα ήθελα να μου πείτε ότι θα ασχοληθεί η Ευρώπη, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε την αίσθηση στην Ισπανία ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και εσείς συγκεκριμένα, ξέρω είχατε κάποιες, ε, κάποιους διαξυφισμούς με την Υπουργού ότι δεν ασχολείται με την τεχνική αρτιότητα των αεροσκαφών η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ιδιαίτερα της Ryanair που κάθε εβδομάδα έχουν προβλήματα και επηρεάζει αυτό και την ασφάλεια. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι η Ryanair είναι αξιόπλοη τέλο πάντων εταιρεία. Ποιο Μαρινέσκου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι είναι μια απαραίτητη πρόταση αυτή. Είμαστε θετικοί. Προσπαθείτε να εναρμονίσετε τα στάνταρ, τα πρότυπα. Αν πρόκειται γι' αυτό, συμφωνούμε. Αλλά δεν θα έπρεπε να συζητήσουμε και το, το να υπάρχει αυτός ο τεχνικός έλεγχος σε όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανεξάρτητα από το που έχει, έχουν εκδοθεί πινακίδες του αυτοκινήτου. No, Καθυστέρησα να βγάλω τα ακουστικά μου γιατί αργούσε η διερμηνία. Θα ήθελα αυτός ο τεχνικός έλεγχος να γίνεται σε όλα τα κράτη-μέλη, ανεξάρτητα από τη χώρα από την οποία προέρχεται το αυτοκίνητο και που, στο οποίο ανήκουν οι πινακίδες. Ο κύριος ε, Ντέχο η κυρία. Είναι απαραίτητη αυτή η πρόταση, δηλαδή να εναρμονίσουμε και τους κανόνες για τον ε, τεχνικό έλεγχο. Ε, επίσης τα περιβαλλοντικά, ένα άλλο σημαντικό θέμα για την ποιότητα των οχήμων. Ε, επίσης ένα σχέδιο ανανέωσης του, του στόλου των αυτοκινήτων γιατί παλιών δεν είναι καλή, καλό. Επίσης, μήπως θα πρέπει να αν αποφασίσουμε ότι απλώς ε, κατεβαίνουν σε... Αν κατέβουν όλα τα αυτοκίνητα σε κυβισμό, δεν θα ήταν πολύ καλό αυτό για το περιβάλλον. Τι θα γίνει επίσης και με, τα, με τις αντίκες να μας πείτε, κύριε Επίτροπε. Δεν ξέρω αν θα σταματήσει τις ε, σκανδαλοθυρικές εφημερίδες να τα βγάζουν αυτά τα θέματα με το λάθος τρόπο, αλλά είναι ένα θέμα που μας απασχολεί. Ένα άλλο σημαντικό θέμα που θέλω να θέσω είναι ότι μπαίνουν, ας πούμε, καμιά φορά ε, λάστιχα στα αυτοκίνητα ε, σε μη τυποποιημένους άξονες. Ξέρετε ότι υπάρχουν ε, οι κυκλικοί άξονες και καμιά φορά και υπάρχουν και άλλου τύπου ε, άξονες, ακτινοτή ας πούμε. Ε, καμιά φορά βάζουμε ε, λάθος λάστιχα σε κυκλικούς άξονες, δηλαδή εκεί πρέπει να βάλουμε λάστιχα σε ακτινοτούς άξονες, θα βάζουμε σε κυκλικούς ας πούμε και δημιουργείται ένα χάος. Ε, επίσης θα πρέπει ε, σε ελέγχου στον δρόμο να τσεκάρουμε ακριβώς το τι είδους λάστιχα έχουν τα αυτοκίνητα και αν είναι ε, τα σωστά λάστιχα για το συγκεκριμένο άξονα. Ε, και επίσης ε, κατά τον έλεγχο στο κταίο ε, θα πρέπει να δούμε αν να τσεκάρουμε συνολικά το αυτοκίνητο. Γιατί δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο συχνά είναι αυτό το φαινόμενο, συνάδελφε. Ένα άλλο σημείο. Χαίρομαι με αυτά που είπε η κυρία Φώστε. Εγώ δεν υποστηρίζω πάντα ότι εμείς θα, πάμε, θα κάνουμε Είμαστε φανταστικοί στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά για την περίπτωση του κταίου μια χαρά τα πάμε. Ε, θέλω μετά από ένα χρονικό διάστημα να έχουμε ετήσιους ελέγχου από επαγγελματίε. Όχι κάθε δύο χρόνια. Αυτό είναι το σωστό, νομίζω. Επίτροπε, έχετε 10 λεπτά και μετά φεύγετε για να προλάβετε και το αεροπλάνο σα. Ευχαριστώ για την υποστήριξή σα στην πρότασή μου. Είμαστε ανοιχτοί σε περαιτέρω συζητήσεις για όλες τις λεπτομέρειες. Να δούμε όλες τις λεπτές αποχρώσεις της πρότασης. Θα τα συζητήσουμε και με ρεαλισμό και με επικοδομητικό πνεύμα. Δεν πρόκειται να δείξουμε ακαμψία. Είμαστε στην αρχική φάση ακόμα. Το είπα και πριν. Δεν θέσατε ερωτήματα όπως αυτά που θέθηκαν κατά τη διάρκεια ε, συνέντευξη τύπου ή από αυτά, σαν και αυτά που με ρώτησε ε, διάφοροι δημοσιογράφοι σε κάποιες χώρες. Ε, με ρώτησαν το γιατί, ας πούμε. Ε, με ρώτησαν αν χρειάζονται μελέτες αντικτύπου. Ξέρετε πολύ καλά ότι όλοι θέλουμε τη μείωση των ατυχημάτων, θανατηφόρων και μη. Αν, υπάρχει, αν όλοι ξέρουμε ότι υπάρχει ένας έλεγχος που, προ, ένας λόγος συγγνώμη, που προκαλεί τέτοιους, τέτοια ατυχήματα θα πρέπει να τον αντιμετωπίσουμε. Ε, με τα τεχνικά πρότυπα και την εφαρμογή τεχνικών προδιαγραφών σε αυτοκίνητα μειώνουμε τα αίτια των ατυχημάτων. Φυσικά, κάθε χώρα μπορεί να πάει παραπέρα, μπορεί να έχει πιο αυστηρούς κανόνες και προϋποθέσεις. Αλλά θέλουμε να εναρμονίσουμε αυτούς τους κανόνες για να έχουμε μια πιο εναρμονισμένη ευρωπαϊκή προσέγγιση. για τις αντίκες. Και εμένα μου αρέσουν οι αντίκες. Μου αρέσουν τα παλιά αυτοκίνητα. Είναι πανέμορφα. Και δεν θεωρούμε ότι μια αντίκα δημιουργεί πρόβλημα στην οδική ασφάλεια. Αν τροποποιηθεί όμως και βάλουμε μια νέα μηχανή, είναι καινούργια από μέσα δηλαδή και απ' έξω αντίκα, τότε νομίζω ότι Πρέπει να το ελέγξουμε αυτό το αυτοκίνητο. Με αυτά τα διαβατήρια των αυτοκινήτων θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα. Ενδιαφέρουσα ιδέα. Για τα περιβαλλοντικά πρότυπα τώρα. Πιστεύουμε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε καλά τέτοια πρότυπα σε ό,τι αφορά την παραγωγή νέων οχημάτων. Έχουμε επίσης περιβαλλοντικούς κανόνες στις τεχνικές προδιαγραφές ε, του αυτοκινήτου, εκπομπές και άλλα τέτοια τεχνικά θέματα. Εδώ ακριβώς μπορούμε να εγγύψουμε και να προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε αυτές τις προδιαγραφές. Για τα λάστιχα που είπε ο Πρόεδρος. Δεν μπορώ να το σχολιάσω. Και για το όριο ταχύτητα. Θυμάμαι ότι όλα όσα έχετε κάνει, ξέρω όλα όσα έχετε κάνει για να αντιμετωπίσετε αυτό το θέμα, το όριο ταχύτητας. Το ζήτημα είναι τι μπορούμε να κάνουμε εμείς. Γιατί αν θεωρείτε ότι το όριο ταχύτητας που υπάρχει ας πούμε στη Γαλλία και το Βέλγιο, αν αυτό το όριο έπρεπε να χρησιμοποιηθεί και στη χώρα μου, θα ήταν τραγικό. Γιατί το όριο ταχύτητα εξαρτάται από την κατάσταση των δρόμων. Και α το αφήσουμε τέλο πάντων, Α αφήσουμε και κάτι στα κρατη να αποφασίσουν. Σε ό,τι αφορά τους παράδρομους, σε ό,τι αφορά το περιθώριο που αφήνουμε ανάμεσα στους μεγάλους δρόμους και στις συνοικίες, ε, τα πεζοδρόμια κτλ. Δεν πρόκειται να πάντως να επιβάλλουμε κανένα ευρωπαϊκό όριο ταχύτητας που θα ισχύει σε όλες τις χώρες. Όχι. Ας το αφήσουμε αυτό στα κράτη-μέλη. Όλα τα κράτη-μέλη έχουν δεσμευτεί να μειώσουν τα τροχέα. Και ένα στοιχείο βέβαια που επηρεάζει τα τροχέα είναι το όριο ταχύτητας. Ανάλογα με τι συνθήκε που υπάρχουν στον δρόμο, λοιπόν, θα πρέπει να προβλέπουμε και το αντίστοιχο όριο ταχύτητα. Α αφήσουμε λοιπόν τα κράτη-μέλη να αποφασίσουν ποιο είναι το ενδεδειγμένο όριο. Κάτι άλλο που ακούστηκε. Αν αγοράσετε ένα αυτοκίνητο. Καταρχάς, είναι δεδομένο θα ξοδέψετε και λεφτά για τα κάψιμα, είναι ένα άλλο θέμα που πρέπει να δούμε, και τους τεχνικούς ελέγχους, εν συνεχεία. Αν κάποιος έχει κάνει ένα προπολογισμό και λέει ότι εγώ θα αγοράσω ένα αυτοκίνητο. Σημαίνει ότι έχει και τα λεφτά για να αγοράσει τη βενζίνη και άρα πρέπει να έχει τα λεφτά και για το κταίο. Ε, τώρα, για το ποιο κάνει τακταίο. Σε ορισμένες χώρες υπάρχουν ιδιωτικές εταιρείε που είναι επιστοποιημένες από τις ε, εθνικές αρχές. Αυτό σημαίνει ότι ελέγχονται από τις εθνικές αρχές αυτές οι ιδιωτικές εταιρείε, ούτως ώστε να σέβονται τις υποχρεώσεις του. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να θεωρούμε μόνο ότι οι δημόσιοι φορείς κάνουν τέτοιους τεχνικούς ελέγχους. Για τις διαφορετικές ε, προδιαγραφές σε διαφορετικές χώρες ε, εκτός Ευρώπης. Έτσι γίνεται συνήθως. Όλες οι χώρες, όπως και η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν τα δικά τους πρότυπα. Εμείς άλλα έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, άλλα έχουν οι Αμερικανοί. Αν θέλουμε να πουλήσουμε αυτοκίνητα στις ΗΠΑ, πρέπει να σεβαστούμε αυτά τα πρότυπα που έχουν εκεί. Γιατί τα αυτοκίνητα που πουλάμε εκεί πρέπει να πληρούν τα δικά τους πρότυπα, τις πολύ αυστηρές προδιαγραφές που έχουν εκεί. Βέβαια και εμείς έχουμε τώρα προδιαγραφές για τα εισαγόμενα αυτοκίνητα. Είναι πολύ λογικό. Ο καθένας που θέλει να εξάγει σε μια αγορά πρέπει να σέβεται τις προδιαγραφές συγκεκριμένη αγοράς. Δεν νομίζω ότι είναι και καινή ώρα για να έχουμε παγκόσμια πρότυπα. Ο στόχος μας είναι να μειώσουμε τα τροχέα πάντως. Μην ξεχνάτε ότι μερικές φορές υπάρχουν πολλές διαφορές ό,τι αφορά τους θανάτους από τροχέα. πούμε, υπάρχει μια χώρα ε, όμορη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει πέντε φορές λιγότερους θανάτους από εμά. Και υπάρχει και μια άλλη, πάλι όμορη και αυτή, τρίτη χώρα, ε, όμορη προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, που έχει τρεις φορές περισσότερα από εμά τροχέα και θανάτους. Ευχαριστώ. Ε, δεν ξέρω αν θα πετάξετε. Με τη Ryanair. Είναι αξιόπλοη η Ryanair. Α, είναι καυτό αυτό το θέμα. Δεν θα αντιδράσω. Μέχρι στιγμή ε, η Ισπανική κυβέρνηση δεν έκανε κανένα αίτημα σχετικά με την Ryanair. Αν ε, υποβάλει σχετικό αίτημα θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για τη Ryanair. Προς το παρόν δεν υπάρχει κανένα αίτημα ισπανικό. Θα είμαστε σε επαφή με την ισπανική κυβέρνηση. Ευχαριστώ πολύ. Καλό σας ταξίδι. Okay, thank you. Next item on the agenda is... Ευχαριστώ πολύ. Το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι οι συμβάσεις παραχωρήσεων και πρόταση του σχεδίου γνωμοδότησης της ε, κυρίας Βίλς. Σαμπίνα, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητοί συνάδελφοι. Τα επόμενα λεπτά θα ήθελα να σας παρουσιάσω το σχέδιο γνωμοδότησης ε, σχετικά με τις συμβάσεις παραχώρησης και να σας εξηγήσω τη θέση μου. Ήδη τον Μάιο του 2010 μεγάλη πλειοψηφία του ε, Κοινοβουλίου υιοθέτησε την ε, πρόταση της Χάιντι Ρούλε. Η έκθεση ήταν ε, κατά μιας νομοθετικής πρότασης της Κομισιόν σχετικά με τις συμβάσεις παραχώρησης παροχής υπηρεσιών δεν πιστεύω ότι υπάρχει καμία ανάγκη για ένα τέτοιο νομοθέτημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ιδιαίτερα φοβάμαι ότι θα υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών και την διασφάλιση της κοινωνικής ασφάλειας. Ως ε, η συγγήτρια της ε, Επιτροπής μας ε, προτείνω να απορρίψουμε το σχέδιο οδηγίας. Να κάνω πρώτα κάποιες γενικές παρατηρήσεις. Βασικός στόχος του σχεδίου είναι η επίτευξη μεγαλύτερου βαθμού ασφαλείας δικαίου. Κατά τη γνώμη μου όμως ε, δεν ε, υπάρχει νομοθετικό κενό. Ούτε μπορούμε να περιμένουμε περισσότερη ε, ασφάλεια δικαίου με την πρόταση αυτή. Η σύναψη συμβάσεως ε, παραχώρηση ρυθμίζεται ε, μέσω του πρωτογενού σε δικαίου Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και ιδίω μέσω των αρχών της ίση μεταχείρισης, της αποφυγή διακρίσεων και της διαφάνειας και μέσω της πάγιας νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Ήδη δηλαδή ρυθμίζεται επαρκώς το θέμα. Επίσης, βρίσκω προβληματική ε, την ασάφεια και την ευρύτητα του πεδίου εφαρμογή στα άρθρα 1, 2 και 5, καθώς και το περιορισμένο εύρο των παρεκκλήσεων στο άρθρο 8. Θεωρώ ότι οι τομεί τη κοινωνική ασφάλιση, του πολιτισμού, τη εκπαίδευση των δημόσιων υποδομών και άλλων δημοτικών υπηρεσιών πρέπει να εξαιρεθούν από το συνολικό πεδίο εφαρμογή. Ε, σημαντική είναι η πτυχή ε, της ε, παροχής υπηρεσιών κοινής ωφελίας. Στο πρωτόκολλο σχετικά με τις υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος τονίζεται το ευρύ περιθώριο δράσης των αρμόδιων δημοσίων αρχών όσον αφορά την παροχή, ανάθεση και χρηματοδότηση υπηρεσιών κοινής ασφαλείας. Στο σχέδιο οδηγίας δεν αναφέρεται σε κανένα σημείο στην ενίσχυση των ε, δημόσιων υπηρεσιών ε, κοινή ωφελία στο πλαίσιο του πρωτογενούς ε, διγέου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι διαπιστώνουμε αντιθέτως. Ε, επιδιώκεται το άνοιγμα του τομέα δημόσιων συμβάσεων στον ανταγωνισμό, αιτιολογικέ σκέψει 1, 2 και 4 και περιορίζεται το, δράση, το περιθώριο δράση για τις αναθέτουσες αρχές, καθώς δεν διαθέτουν απεριόριστη ελευθερία επιλογής κατά τον καθορισμό των κριτηρίων ανάθεσης. Ως ε, συνδικαλίστρια, ε, επικρίνω ιδιαίτερα ότι δεν προβλέπεται η τήρηση των τοπικών συλλογικών συμβάσεων κατά την ανάθεση δημοσίων ε, συμβάσεων. Επίσης, ε, η Επιτροπή επικεντρώνεται στη ε, δημιουργία νέων ε, τομέων της αγοράς, αντί για την διασφάλιση κάποιων υπηρεσιών κοινή ωφελία. Οι υπηρεσίες αυτές καλύπτουν κάποιες βασικές ανάγκες των ανθρώπων και δεν επιτρέπεται να υπόγειται στις αρχές της αγοράς. Του ε, θέλουμε ποιοτικές ε, και ε, γενικές υπηρεσίες που να παρέχονται παντού. Φοβάμαι ότι οι συμπράξεις δημοσίου, δημοσίου, δημοσίου τομέα θα αποτελούν εξαίρεση. γενικά με το σχέδιο προβλέπεται καλύτερη πρόσβαση στην αγορά για τις επιχειρήσεις και η προώθηση των συμπράξεων δημόσιο-ιδιωτικού τομέα. Ε, ε, είναι αυταπάτη να πιστεύουμε ότι ε, θα έχουμε μεγαλύτερη διαφάνεια και αποτελεσματικότητα καθώς και χαμηλότερο κόστος. Όσον αφορά τον τομέα των μεταφορών, διαπιστώνουμε ότι η προτινόμενη οδηγία όσον αφορά τις μεταφορές, τις σιδηροδρομικές μεταφορές, τα τραμ, τα λεωφορεία, ή τα τρόλεϊ ε, κλπ. θα ακολουθήσουν και ε, τον δρόμο των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Προβλέπετε Η προτινόμενη οδηγία ισχύει και για, τις, ε, για την ναυσιπλοεία, την εσωτερική ναυσιπλοεία ε, και άλλους μεταφορείς. Υπάρχει ο κανονισμός 1008 ε, και κάθετος 2008 καθώς ε, και, ε, καθώς και το νομοθέτημα 1370 κάθετος 2007. Ε, Πιστεύω ότι δεν χρειαζόμαστε ειδική ρύθμιση για τις συμβάσεις παραχώρησης. Η πρόταση της Κομισιόν δεν θα οδηγήσει σε βελτίωση της παρούσας κατάστασης. Του αντίον θα προκαλέξει σύγχυση σε σχέση με τους ισχύοντες κανόνες. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Από το ΕΛΚ, ο κύριος Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ και την εισηγήτρια ε, για την ανάλυση της. Είναι γεγονός ότι απαραίτητο σε μια εσωτερική αγορά όπως είναι η ευρωπαϊκή αγορά ε, να υπάρχει ε, έτσι ανταγωνιστικότητα, να τονώνεται ο ανταγωνισμός και η ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών. Συμφωνούμε γι' αυτό. Και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά ε, στις συμβάσεις παραχώρησης να υπάρχει τέτοια δυνατότητα υπό όρους. Μα έχουμε αρκετούς νόμους και πολλούς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει τώρα μια πρόταση για να τα συγκεκριμενοποιήσει όλα αυτά και να τα διευκρινίσει. Πιστεύω ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε μια διάκριση ανάμεσα στις ΔΕΚΟ, ε, του δημοσίου δηλαδή, και στις ιδιωτικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών οι κρίσιμες υποδομές όπως είναι δίκτυα ε, παροχής ενέργειας ή η φαρμακευτική περίθαλψη, η υδροδότηση, η αποχέτευση. Όλα αυτά θα πρέπει να τα συζητήσουμε όταν συζητάμε για τα θέματα της ιδιωτικοποίησης και της απελευθέρωσης αγοράς στη Γερμανία ε, και στη Γερμανία όπως πήγαν τα πράγματα τα τελευταία χρόνια δεν είναι συνταρακτικά. Ε, στην αρχή ωρεοποιούν, ας πούμε, μειώνεται ε, το νερό και αποχέτευση ε, για διαφήμιση και μετά όταν έχουν ε, συμπολογίσει όλο το κόστος και την εξυγίαση και τα λοιπά, το δικτύο αυξάνονται μέχρι και 60% και η ίδρυυση και η αποχέτευση. ε, των διακρίσεων σωστό, όταν υπάρχει δυνατότητα δημόσιας ανάθεσης για όλους αλλά με συγκεκριμένες προϋποθέσεις έτσι, για τις εταιρείες που υποβάλλουν, ε, ε, ε, εκδηλώνουν ενδιαφέρον. Γι' αυτό καταρχήν συμφωνούμε, μεν, αλλά να μην ανοίξουμε ακόμα περισσότερο τους ασκούς του αιώλου. Επίσης η αρχή της αμοιβαιότητας είναι το πιο σημαντικό. Αμοιβαιότητα. Πρόκειται για την ευρωπαϊκή αγορά και για κοινοφιλείς υπηρεσίες σε διάφορα κράτη-μέλη. Στις μεταφορές νομίζω ότι είναι καλή η πρακτική που επικρατεί. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το πακέτο των σιδηροδρόμων και την αναδιατύπωση και ε, στην εθνική ε, νομοθεσία ακριβώς για το σιδηρόδρομο. Θα πρέπει να ανοίξει περισσότερο αυτή η παροχή υπηρεσιών για τους ε, πολίτες και τους επιβάτες. Αυτό μπορεί να γίνει και στη θάλασσα και στον αέρα, όχι μόνο στην ξηρά. Δεν χωρά καμία αμφιβολία. Αλλά για τις ε, κοινοφελείς υπηρεσίες και τις ε, καινοτομίες να το ξανασυζητήσουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ο Σάιντ Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την εισαγωγή της. Ε, ε, εξέφρασε και μια σειρά επικρίσεων στην πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πρέπει να πω ότι σε μεγάλο βαθμό συμφωνούμε μαζί της. Πλην όμως δεν έχουμε πιστεί ακόμα από το γεγονός ότι η πρόταση ε, θα πρέπει να απορριφθεί απλούστατα. Θα τα δούμε τις επόμενες μέρες, ε, να τα μελετήσουμε μήπως μπορούμε να βελτιώσουμε την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συγκεκριμένα ε, στους λιμένες. Ε, νομίζω θα είχε μεγαλύτερο νόημα να ε, υπάρξει κάποια ρύθμιση και να μην τα απορρίψουμε συλλήβδη. Λοιπόν, θα το ξανακοιτάξουμε. Πάντως συμφωνούμε ότι η αφετηρία χρειάζεται έτσι μια κριτική ματιά. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Οζίας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε Σίμψον. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω και την εισηγήτρια κυρία Βίλς για το έργο της, αλλά κατανοώ τις ανησυχίες της, αλλά δεν συμμερίζομαι το αίτημα της απόρριψης της πρότασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πιστεύω αντιθέτως ότι η νομοθετική πρωτοβουλία για τις παραχωρήσεις είναι ε, αναγκαία για να μην πω απαραίτητη και χρήσιμη για να έχουμε ένα νομοθετικό πλαίσιο. Και, ε, ε, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις δημόσιες συμβάσεις. μέχρι τώρα έχουμε και αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστήριου λαμβάνουν θέση διάφοροι, ε, ε, προσφεύγουν στο δικαστήριο, έχουμε πολλές αποφάσεις. Αυτό σημαίνει ότι είναι ε, πάρα πολύ ασαφής η νομοθεσία και θα πρέπει να επέμβει ο νομοθέτης για να επανέλθει ασφάλεια δικαίου. Για το λόγο αυτό λοιπόν είμαστε τώρα σε ένα σταυροδρόμι και χρειαζόμαστε ένα κείμενο ρυθμιστικό που θα περιορίζει τις νομικές ασάφειες. Η πρόταση της Κομισιόν είναι ένα καλό σημείο θετηρία προς αυτήν την κατεύθυνση. Οφείλω να πω ότι το κείμενο παρόλα αυτά μου φαίνεται υπερβολικά δύσκολο, έχει πολλές διατυπώσεις και αναφέρεται πολλές οι διαδικασίες. Θα πρέπει να γίνει μια προσπάθεια απλούστευσης της οδηγίας. Ακριβώς για να έχουμε ένα χρήσιμο εργαλείο, απλό για τους ενδιαφερόμενους και να έχουμε ένα σαφέστερο πιο ρεαλιστικό και πιο αποτελεσματικό πλαίσιο. Διαφορετικά από ό,τι λέει η συγγήτρια, εγώ θεωρώ ότι περιορίζεται η διακριτική δυνατότητα της, ε, των αρχών. Δεν ε, αυξάνεται. Πρέπει να πούμε επίσης ότι πρέπει να υπάρχει μια κάποια ευελιξία για να υπάρχει έτσι ένα περιθώριο ελευθερίας. Γιατί με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται υψηλή, υψηλές υπηρεσίες για τους ε, πολίτες ε, που είναι σημαντικό για αυτές τις υπηρεσίες. Άκουσα από τους εισηγητές να αναφέρονται σε διαφορετικές διατάξεις. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να διευκρινίσουμε καλύτερα τα περιθώρια εφαρμογής της οδηγίας. Ε, γιατί έγιναν κάποιες διευκρινήσεις στην αιτιολογική σκέψη ε, θα πρέπει να αποκλείσουμε σαφέστατα κάποιες ε, παραπομπές, παραδείγματο χάρη, στις υπηρεσίες ε, που παρέχονται στις ακτές, ας πούμε, που, που δημιουργούν τόσα πολλά προβλήματα σε πολλές εθνικές νομοθεσίες, παραδείγματο χάρη στην, στην Ιταλία, λόγω της ιδιαιτερότητας του τουριστικού τομέα. Είναι σημαντικό επίσης η... οι αρμοδιότητες που δίνουμε σε ορισμένες δημόσιες αρχές και, στις, και σε εταιρείε που συνδέονται με αυτές. Αυτά. Ο κύριος Ντεμπάκερ. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ και την εισηγητρία για την εισαγωγή της στη συζήτηση. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό που προτείνει. Λαμβάνει μια νομοθετική πρωτοβουλία Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να διαλύσει αυτή την ασάφεια που υπάρχει. Είναι πολύ τόσο απαραίτητο γιατί είναι πολύ περίπλοκη η κατάσταση και με τις παραχωρήσεις. Ε, θέλει μεγαλύτερη διαφάνεια, η συμμεταχείριση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτό είναι περισσότερο απαραίτητο από ε, ποτέ, γιατί δραστηριοποιούνται όλο και περισσότεροι επιχειρηματίε σε αυτό το κλάδο. Η πρόταση έχει προστιθέμενη αμυναξία, Βεβαίως χρειάζονται αλλαγέ να γίνουν στην πρόταση αυτή ε, και χωράει και συζήτηση. Αλλά απόρριψη, η συλλήφθη νομίζω είναι κακή ιδέα. Σε ένα συγκεκριμένο θέμα θέλω να αναφερθώ και να μιλήσω για τους λιμενικούς ε, ε, το, τις λιμενικές υπηρεσίες και τον τομέα των λιμένων γενικά είναι εμπίπτη στην εγκάρση αυτή η οδηγία και θα πρέπει να κοιτάξουμε ε, να έχουμε μια πιο στοχευμένη και ειδική προσέγγιση γιατί έχουμε ε, ε, leasing, παραχωρήσεις, εκχωρήσεις και μια σειρά άλλων πραγμάτων στα λιμάνια και είναι κάτι το οποίο χρειάζεται ξεχωριστή μεταχείριση και να το δούμε αυτό στην επόμενη συζήτηση. Thank you very much for the commission. It's... Ευχαριστώ από την Κομισιόν. Ευχαριστώ και τον εισηγητή για το σχέδιο έκθεσης. Ευχαριστώ για όλα τα σχόλια που ακούσαμε κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Να σχολιάσω αυτά που ακούσαμε λίγο και σα λέω βεβαίω ότι είναι στη διάθεσή της Κομισιόν για περαιτέρω συζητήσει και λεπτομέρειε. Καταρχά να τονίσω ότι η πρόταση έχει σαν σκοπό να αντιμετωπίσει περίπλοκα θέματα σε ό,τι αφορά τις συμβάσεις παραχώρησης που είναι μακροχρόνιες και έχουν την τάση να δημιουργούν πρόβλημα στην αγορά αν εφαρμόζονται με λάθος τρόπο. Ε, θέλαμε δηλαδή ε, τη χρόνια έλλειψη διαφθοράς ε, στην νέα αγορά να την αντιμετωπίσουμε για τις δημόσιες συμβάσεις. Και σε ό,τι αφορά τις συμβάσει συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών, στις υπηρεσίες, αυτό δεν υπάρχει σήμερα. Ε, θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που ήδη υπάρχουν. Ε, το σχέδιο οδηγία, 62 θέλει να δώσει μεγαλύτερη ασφάλεια στις ε, δημόσιες αρχές όταν δίνουν τέτοιε παραχωρήσει, ούτω ώστε ε, να είμαστε σίγουροι ότι ο τρόπος παραχώρησης, ε, ο τρόπος παραχώρησης αυτής της σύμβασης έχει γίνει με το σωστό τρόπο, Ούτω ώστε να μην υπάρχει ζημία ούτε για του επιχειρηματίε ούτε για τι δημόσιε αρχέ. Αλλά η πρόταση αυτή, και θέλω να το ξεκαθαρίσω, δεν αφορά, δεν αφορά την ιδιωτικοποίηση κάποιων ε, υπηρεσιών. Έχει συζητηθεί πολύ αυτό το θέμα στην Επιτροπή ΙΜΚΟ και μία από τις προτάσεις στην έκθεση του εισηγητή είναι να διευκρινίσουμε πάρα πολύ αυτό το σημείο. Όμως το κείμενο της Κομισιόν δεν, δεν ήταν να μιλήσουμε για την ε, ιδιωτικοποίηση ή εξωτερήκευση των υπηρεσιών. Όχι, θέλουμε να δώσουμε τη δυνατότητα στι δημόσιε αρχέ. Αν αποφασίσουν να κοιτάξουν ένα πάροχο υπηρεσιών και να το βρουν στην αγορά, να το κάνουν μέσα σε ένα πλαίσιο ασφαλεία δικαίου. Μια σύντομη αναφορά σε δύο σημαντικέ δηλώσει που ακούστηκαν κατά τη διάρκεια τη συζήτηση. Ε, για τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος. Να επαναλάβω ότι είπε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ότι οι υπηρεσίες της διασφύσης καλύπτονται επίσης από τους κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις και τις παραχωρήσεις. Δεν υπάρχουν ε, εξαιρέσεις εδώ σε αυτές οι υπηρεσίες. Καλύπτονται επίσης ε, με βάση την νομοθεσία, την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Δεύτερον, για το κατά πόσο αντιμετωπίζει πλήρω το ΔΕΚ την ομολογία του τη συμβάση παραχώρησης. Στα δέκα, τελευταία χρόνια το δικαστήριο ε, εξέδωσε 26 αποφάσεις. Δεν μπορείτε να πείτε ότι δεν είναι ξεκάθαρες οι φάσεις της διαδικασίας. Και επίσης ο ρόλος του συνομοθέτη είναι, δηλαδή του του, των κρατών μελών και, το και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι πάρα πολύ σημαντική ε, για να ξεκαθαρίζει σημεία που δεν έχουν ξεκαθαρίσει το δικαστήριο ε, με την ομολογία του. Ε, τώρα, για το ποιος είναι καλύτερος πάροχος υπηρεσιών, κάποια εταιρεία ή κάποια δημόσια αρχή. Εμείς είμαστε ουδέτεροι προς αυτό. Θέλουμε να έχει πρόσβαση όποιος το επιθυμεί και την απόφαση την παίρνουν οι δημόσιες αρχές. Δεν είναι υποχρεωτικό να χρησιμοποιήσουν αυτούς τους παρόχους υπηρεσιών. Είναι μια δυνατότητα και απλώς θέλουμε να έχουμε ένα ασφαλές πλαίσιο εκχώρησης αυτών των συμβάσεων. Τίποτε άλλο. Αυτή η συζήτηση είναι πολύ λεπτή, πολύ ευαίσθητη και έχει γίνει για πολλά χρόνια. Η Επιτροπή ΙΜΚΟ ε, ζήτησε να γίνουν τρεις επιπλέον μελέτες ε, για, σχετικά με την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Και έχουμε καταλάβει ότι υπάρχει ένα πρόβλημα στην αγορά. Ε, πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε αυτές τις ελλείψεις για να είναι σε καλύτερη θέση και οι δημόσιες αρχές που αναζητούν ε, ιδιωτικούς παρόχους αλλά και οι εταιρείε. Είμαστε στη διάθεσή σας να κοιτάξουμε περαιτέρω το κείμενο και αν μπορούμε να βελτιώσουμε οτιδήποτε, κανένα πρόβλημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Wills, θέλετε να απαντήσετε. Ναι. Ήθελα να ευχαριστήσω καταρχήν όλους τους σκιώδεις εισηγητές και τους άλλους ομιλητές για τις παρατηρήσεις τους και τη συμβολή τους στη συζήτηση. Νομίζω ότι ο κύριος Κούν κατέστησε σαφές Ποιος είναι ο ιδιαίτερος ε, ρόλος ε, των ε, υπηρεσιών κοινή ωφελίας. Πρόκειται για υπηρεσίες τις οποίες χρειάζονται οι πολίτες και πιστεύω ότι οι υπηρεσίες κοινή ωφελία. δεν θα πρέπει να υπόκεινται στους κανόνες της αγοράς και του κέρδους φυσικά. τα ε, οι Δήμοι μπορούν να ε, κάνουν κοινοπραξίες δημοσίου-δημοσίου ε, και να οργανώσουν από κοινού τις υπηρεσίες αυτές. Δεν βλέπω όμως να υπάρχει καμία ανάγκη να ανοίξουμε στην αγορά την πόρτα προς τις υπηρεσίες κοινής ωφελίας. Οι συμπράξεις ιδιωτικού και δημοσίου τομέα ε, όπως λέει η Κομισιόν, ε, δεν νομίζουμε ότι θα προωθήσουν τις υπηρεσίες αυτής. Ε, εγώ ε, από τον Βούργο προέρχομαι και είδαμε τέτοιες ε, συμπράξεις. Εκεί είδαμε ότι οι ιδιώτες, ε, ο ιδιωτικό τομέας όταν θέλει να συμμετάσχει εκεί θέλει να λάβει και κέρδος, άρα αυξάνεται το κέρδος. Για παράδειγμα στο χτίσιμο σχολείων πια δεν υπάρχει ευελιξία όσον αφορά τις συμβάσεις αυτής, διότι οι συμβάσεις αυτές δεν είναι ευέλικτες επειδή έχουν μεγάλη διάρκεια ε, συχνά 40 χρόνια ή κάτι τέτοιο και ε, η Κομισιόν το αναφέρει αυτό και ε, χάνεται ευελιξία αν έχουμε τέτοιες συμπράξεις και όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις υπάρχει επικάλυψη με τον τομέα των οικοδομών και δεν πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρξει περισσότερη ρύθμιση για τους λιμένες. Ε, μας απείλησαν με ένα πακέτο λιμένων υπαριθμών 3, αλλά μας ενδιαφέρει περισσότερο, ε, να μην υπάρχουν συμβάσεις παραχώρησης ε, για ε, τα οικόπεδα. Δεν χρειάζεται σύμβαση παραχώρησης για, την, για τις άλλες δουλειές του λιμένα. Πρόκειται λοιπόν για άλλη κατάσταση. Επίσης, τροπιαστικό στην πρότασή της Κομισιόν βρίσκω το ότι η υπάρχει δέσμευση όσον αφορά τα κριτήρια κατά την ανάθεση ε, και ότι κάποια κριτήρια δεν μπορεί να τα απαιτήσει κανείς από τον ιδιωτικό τομέα. Εάν ε, ζητάει κανείς από ε, ιδιωτική επιχείρηση δεν δεσμεύεται να συμμετάσχει, δεν δεσμεύεται αυτή από τις συλλογικές συμβάσεις, ενώ μια δημόσια σύμβαση, αν ε, θέλει να συμμετάσχει, ε, κρίνεται μόνο με βάση το, ε, την τιμή. Υπάρχουν λοιπόν πολλά επιχειρήματα να απορρίψουμε αυτή την πρόταση οδηγίας. Όπως άλλωστε πρόκειταν και άλλοι συνάδελφοι από άλλες επιτροπές. Μπορούμε να συνεχίσουμε τις συζητήσεις, να συναντηθούμε με τους εσκιώδεις εισηγητές και πιστεύω ότι έτσι θα μπορέσουμε να βρούμε έναν τρόπο να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου μπορείτε να καταθέσετε τροπολογίες. Θα ψηφίσετε στην Επιτροπή Μεταφορών στις 6 Νοεμβρίου, στην Επιτροπή ΙΜΚΟ στις 18 Δεκεμβρίου. 27 Σεπτεμβρίου για σας λοιπόν, για να καταθέσετε α, τροπολογίες. 6 Νοεμβρίου ψηφίζουμε. 18 Δεκεμβρίου ψηφίζει ΙΜΚΟ. Πολύ ωραία. Περιμένω τώρα τους συντονιστές και σταματώ εδώ τη συνεδρίαση. Παρακαλώ να μαζευτούν οι συντονιστές το συντομότερο δυνατόν.